Γεια σας, σας καλωσορίζω. Βιαστήκαμε όλοι να γυρίσουμε εδώ. Χαίρομαι πάντως που έχουμε μαζί μας και τον Επίτροπο Μπαρνιέ και τον Επίτροπο Αλμούνια για αυτή τη δημόσια ακρόαση και θα ήθελα να καλωσορίσω όλους τους ομιλητές. Με την ακρόαση αυτή θέλουμε να συνεισφέρουμε στη συζήτηση για τις ε, κρατικές βοήθειες που έχουν σαν στόχο να στηρίξουν την οικονομία κατά τη διάρκεια της ε, κρίσης η οποία εξακολουθεί να σοβεί και να εξετάσουμε επίσης και τις στρατηγικές εξόδου από τα προγράμματα που αποφασίσαμε στο τέλος του 2008 σχετικά με την υποστήριξη του χρηματοπιστωτικού τομέα κατά τη διάρκεια της κρίσης. Θα υπάρξει συνέχεια μετά την ακρόαση αυτή, θα υπάρξει η δυνατότητα να κατατεθούν τροπολογίες στην έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού του 2009, την οποία προετοιμάζει ο Έπινγκ. Και αλλάζουμε και τον τίτλο της έκθεσης αυτής, αναθεώρηση των ενδιάμεσων μέτρων κρατικών βοηθειών για την αντιμετώπιση της κρίσης. Η προθεσμία για τις τροπολογίες αυτές είναι η 7η Οκτωβρίου πέμπτη απογευματινή. Θα υπάρξουν δύο πάνελ. Στο πρώτο θα είναι με τους δύο επιτρόπους. Θα συγκεντρώσουν στην προσοχή τους τα μέτρα τα οποία έχει προτείνει και έχει λάβει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ένα δεύτερο πάνελ θα αποτελείται από εμπειρογνώμονες και την απάντηση της αγοράς. Στο πρώτο πάνελ κάθε επίτροπος έχει 10 λεπτά, θα ακολουθηθούν ερωτήσεις από πλευράς των μελών και το δεύτερο πάνελ, κάθε ομιλητής θα έχει 5 λεπτά και θα ακολουθήσει η, θα ακολουθήσει η περίοδος των ερωτήσεων. Έχουμε ταυτόχρονη διερμηνία όπως έχετε ίσως διαπιστώσει, δεν χρειάζεται όμως να βιάζεστε πάρα πολύ για να χωρέσετε περισσότερα πράγματα μέσα στα 5 ή στα 10 λεπτά. Ε, έχουν διανεμηθεί επίσης και τα βιογραφικά των ομιλητών και θυμίζω ότι αναμεταδίδεται δικτυακά η συνεδρίαση αυτή και ε, μας ακούν και μας βλέπουν σε πραγματικό χρόνο. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα ήθελα να ξεκινήσω δίνοντας το λόγο στον Επίτροπο Αλμούνια για 10 λεπτά. Ελπίζω να είστε γενναιόδωρος μαζί μου, αν πάρω λίγα περισσότερα από τα 10 λεπτά, λόγω όλων αυτών που έχουν συμβεί τα τελευταία δυόμιση χρόνια. Θα ήθελα λοιπόν, σε αυτά τα 12 λεπτά με την άδειά σας, να σας μεταφέρω ε, τα εξής. Να σας πω τι έχουμε κάνει από τότε που ε, έκλεισε η εταιρεία Λίμαν μέχρι σήμερα στον τομέα της βοήθειας, στον τομέα των χρηματοπιστωτικών και στον ευρύτερο τομέα. Σχετικά με τον χρηματοπιστωτικό τομέα για πρώτη φορά χρησιμοποιήσαμε από τον Οκτώβριο του 2008, αμέσως μετά δηλαδή την πτώχευση της Λίμαν, το άρθρο 107β, 3β. Είναι η έκτακτη νομική βάση η οποία θα χρησιμοποιείται σε έκτακτες περιπτώσεις. Βλέπετε ότι χρησιμοποιώ συνεχώς τη λέξη έκτακτος. Η νομική αυτή βάση χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά λοιπόν στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε η συνθήκη της Ρώμης, προσπαθούμε να ενισχύσουμε το σύνολο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, γιατί αντιμετωπίζει έναν λεγόμενο συστημικό ακριβώς κίνδυνο, και έχει επηρεάσει φυσικά και το σύνολο της οικονομίας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει χρησιμοποιήσει τις έκτακτες δυνατότητες που δίνει η βάση 107.3 με τέσσερις ανακοινώσεις τον Οκτώβριο του 2008 για τα πιστοτικά ιδρύματα και για την εσωτερική αγορά. Το Δεκέμβριο του 2008 μια δεύτερη ε, ανακοίνωση για την ισροή κεφαλαίων στα πιστοτικά ιδρύματα για να αποκαταστήσουμε δηλαδή τις συνθήκες, να περιορίσουμε τις συμβατές βοήθειες και παρεμβάσεις σε αποδεικτά επίπεδα και να αποφύγουμε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού. Το Φεβρουάριο του 2009 the restructuring communication Υπήρξε η ανακοίνωση για τα μέτρα αναδιάρθρωσης αυτό τον Ιούλιο του 2009. Τι θέλουμε τελικά να πετύχουμε με όλα αυτά τα πακέτα των έκτακτων γενικά μέτρων τα οποία πήραμε. Καταρχάς αυτό που θέλουμε να πετύχουμε είναι η ε, χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Δεύτερον θέλουμε να, έχουμε, ε, ε, να μην υπάρχουν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό και να μην υπάρξει μια πολυδιάσπαση της εσωτερικής αγοράς και να μην υπάρχουν βαθύτερες διαφοροποιήσεις στον τομέα αυτό και θέλουμε επίσης να προχωρήσουμε και στην αναδιάρθρωση των θεσμικών οργάνων τα οποία θεωρούμε ότι, ε, ε, ότι χρειάζονται ε, βοήθεια για να μπορέσουν να ξεφύγουν από την κρίση και να καταλήξουμε εκ νέου σε ένα ανταγωνιστικό υγιές πιστοτικό σύστημα. Οι κυβερνήσεις ανέλαβαν την υποχρέωση από τον Οκτώβριο του 2008 μέχρι τον Αύγουστο του 2010 καταλήξαμε σε 4-3 που είναι περίπου το 39% του κοινοτικού ΑΕΠ, 30% σε επίπεδο κρατικών εμπειρήσεων, 4,45% με ενέσεις κεφαλαίου, και μικρότερα επίσης μικρότερα ποσά για απομειωμένα περιουσιακά στοιχεία. Από τον Οκτώβριο του 2008 μέχρι τον Αύγουστο του 2009 έχουμε, έχουν περιπτώσει και σαν ένωση και σαν χώρες ε, περίπου δώσει άλλο ένα 17% του κοινοτικού ΑΕΠ κάτω δηλαδή του μισού από αυτά τα οποία είχαμε αναλάβει στο παρελθόν. Ε, that ε, were 15 for... 15 λοιπόν προγράμματα ε, για τις ενέσεις κεφαλαίου που εξακολουθούν να λειτουργούν πολλές από αυτές, οκτώ θα είναι γιατί από ό,τι ακούσαμε η Φιλανδία θα διακόψει τα προγράμματά της αυτά στο τέλος του μήνα δύο επίσης ε, προγράμματα δεσμεύσεων για την Γερμανία και την Ιρλανδία για απομειωμένα ε, περιουσιακά στοιχεία, έξι προγράμματα για την διασφάλιση ρευστότητας πιστοτικών ιδρυμάτων, πέντε από αυτά λειτουργούν ακόμα και 21 προγράμματα εγγυήσεων από τα οποία τα 12 έχει παραταθεί η λειτουργία τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2010 και σε 12 χώρες είναι πολύ πιθανό να ζητηθεί να παραταθούν αυτά τα προγράμματα εγγυήσεων στο μέλλον. Έχουν υπέρξει επίσης σχετικά με τις εθνικές αποφάσεις ε, γύρω από 44 περιπτώσεις κρατικών παρεμβάσεων έχουν ε, εξεταστεί 27 οι οποίες έχουν κλείσει και έχει ληφθεί τελική απόφαση. Στις 23 από τις 27 η απόφαση και η κρίση, η αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν θετική ε, σε τρεις περιπτώσεις υπήρξε πτώχευση ε, του Ιδρύματος και σε μία περίπτωση η απόφαση ήταν αρνητική και ζητήθηκε να ε, πάρουν πίσω τα χρήματα που έδωσε το Πορτογαλικό Δημόσιο. Και σε 17 περιπτώσεις συνεχίζεται η αξιολόγηση και εξετάζουμε λοιπόν αυτές τις περιπτώσεις οι οποίες συνολικά επαναλαμβάνω σήμερα είναι 27. Εγώ τώρα προσπαθώ να σας παρουσιάσω συνολικά τα προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να αναλύσουμε. Έχουμε την Ιρλανδική περίπτωση, δεν θα επιμείνω πάρα πολύ στην Ιρλανδική περίπτωση, γνωρίζετε την κατάσταση, έχουμε την Ελληνική περίπτωση, και ξέρετε ότι έχουμε και το ε, μεικτό πρόγραμμα χρηματοδότησης της Ελλάδας εδώ και λίγους μήνες, ε, μεικτό εννοώ ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ένα ταμείο σταθερότητας 10 δις, το οποίο συνδέεται άμεσα με τις δυνατότητες ε, βοήθειας των τραπεζών εφόσον το χρειάζονται στην Ελλάδα. Έχουμε επίσης τα προβλήματα τα γερμανικά, τις Landesbanken, Ήδη ε, εξετάζουμε τρεις τέτοιες περιπτώσεις. Σε δύο από αυτές τις περιπτώσεις έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολύ δύσκολες συζητήσεις πριν καταλήξουμε στην τελική απόφαση για την αναδιάφθρωση μεταρρύθμιση αυτών των πιστοτικών ιδρυμάτων και έχουμε επίσης και την περίπτωση ε, της ε, HIPO Estate, Estate που έχει ένα πρόβλημα ενεργητικού άνω του 1,7 δις. Και στο μέλλον θα αντιμετωπίσουμε και άλλες τέτοιες περιπτώσεις σχετικά με ορισμένα πιστοτικά ιδρύματα τα οποία θα χρειαστεί να, δώσουμε, να ζητήσουμε να υπάρξουν νέα χρήματα από πλευράς ε, της, ε, του δημοσίου είτε είναι στην Ισπανία είτε σε άλλες χώρες Έχουμε λοιπόν πολλή δουλειά η οποία συνεχίζεται. Η ανανέωση του οικονομικού αυτού πακέτου προσπαθούμε να δούμε πώς θα προσαρμόσουμε μία από αυτές τις τέσσερις ε, ανακοινώσεις οι οποίες αναφέρθηκαν από μένα προηγουμένως ε, αυτή που αφορά την αναδιάρθρωση που θα λήξει στο τέλος του 2010, εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξουν εξέκτακτες ρυθμίσεις σχετικά με την αναδιάρθρωση των πιστοτικών ιδρυμάτων και για το 2011, αλλά όχι όμως κάτω από τις ίδιες συνθήκες και προϋποθέσεις που κάτι τέτοιο ισχύει φέτος. Θα πρέπει να σκληρύνουν οι προϋποθέσεις αυτές. Θα θέλαμε σαν παράδειγμα ήδη από του χρόνου να ζητήσουμε να υπάρξουν αξιολογήσεις για τη βιωσιμότητα όλων των πιστοτικών ιδρυμάτων στα οποία επενδύεται δημόσιο χρήμα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν την προοδευτική σταδιακή αν θέλετε αποχώρηση από όλους αυτούς τους τομείς των παρεμβάσεων ε, με εξαίρεση ίσως το θέμα των εγγυήσεων και ε, φυσικά θα σκληρύνουμε και τις προϋποθέσεις για τη μεταρρύθμιση αναδιάφρωση των πιστοτικών ιδρυμάτων. Ζήτησα από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ξεκινήσουν ε, ε, επίσης για τη διατύπωση των κατευθυντήριων γραμμών των ιδρυμάτων αυτών ή ιδρυμάτων πιστοτικών κάτω από κανονικές συνθήκες και θα ήθελα οι κατευθυντήριες γραμμές αυτές να είναι ήδη έτοιμες από το 2012 σχετικά με το ε, μη χρηματοπιστωτικό τομέα της οικονομίας μας. Ξέρετε ότι πήραμε κάποια μέτρα ήδη από τον Οκτώβριο του 2008, νέες βοήθειες, ε, επιτρέπεται 400.000 ε, να πηγαίνουν χωρίς συγκεκριμένη αδειοδότηση μέχρι το ποσό αυτό και επίσης και σε επίπεδο ε, ασφάλειας ε, για ε, τις εξαγωγές. Έχουμε επίσης επιτρέψει συνολικά 80, 81 τέτοιες περιπτώσεις επιδότησης του τομέα του μη πιστοτικού τραπεζικού. 23 από αυτές είναι χωρίς προϋποθέσεις γιατί είναι κάτω από ένα συγκεκριμένο ποσό Έχουμε επίσης αντιμετωπίσει και την περίπτωση, πέντε μάλλον περιπτώσεις για τη μείωση του επιτοκίου για χρηματοδότηση λεγόμενων πράσινων προγραμμάτων και υπάρχουν και άλλου είδους ε, κατηγορίες. Από τον Οκτώβριο του 2008 ε, μέχρι τον Απρίλιο του 2010 που είναι η τελευταία τελική αριθμή τους οποίους έχω, έχουμε αδειοδοτήσει προγράμματα και δεσμεύσεις 185 δις από τις 27 χώρες, αλλά έχουμε πάρει πληροφορίες για την πληρωμή μόνο 21 δις από τα 185 τα οποία, για τα οποία είχαν δεσμευθεί οι χώρες. Προχωρούμε τώρα στο phasing out, στη στανδιακή αποχώρηση αυτής της διαδικασίας από το τέλος του 2010 ε, δεν είμαστε απόλυτα σε θέση βέβαια να καταργήσουμε πλήρως αυτό το προσωρινό ρυθμιστικό πλαίσιο σε όλο τον κόσμο και όλα τα μέσα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας. Εξακολουθούν κάποια από αυτά και χρειάζονται. Πιστεύω και πρότεινα ήδη στα κράτη-μέλη η δυνατότητα των 500.000 να καταργηθεί στο τέλος του χρόνου, αλλά παρόλα αυτά κάποια μέτρα θα πρέπει να ισχύσουν και το 2011 και να γίνουν λίγο πιο αυστηρά σχετικά με τις επιδοτήσεις των εγγυήσεων και των δανείων. Ίσως επίσης να παραταθούν και οι επιδοτήσεις για τα πράσινα προϊόντα και τα πράσινα προγράμματα που έχουν χρησιμοποιηθεί σε ελάχιστα κράτη-μέλη. Λίγες είναι οι χώρες που έχουν χρησιμοποιήσει αυτή τη δυνατότητα, παρότι τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στο συγκεκριμένο τομέα είναι παρόμοιες σε όλες τις χώρες. Και τελειώνω εδώ πρόεδρε, πιστεύω ότι θα πρέπει να προτείνουμε προς τα κράτη-μέλη και θα ήθελα και ε, κάποια ενημέρωση από πλευράς τους να μετασχηματίσουμε σε μόνιμη κατευθυντήρια γραμμή ε, βοήθειας ε, τις προϋποθέσεις για τα risk capitals όπως επίσης και την ασφάλεια για τις επιδοτήσεις της εξαγωγές. Βλέπουμε λοιπόν ότι χρησιμοποίηθαν τεράστιες, τεράστια ποσά από το δημόσιο χρήμα, κυρίως χρησιμοποιήθηκαν τα ποσά αυτά στον χρηματοπιστωτικό τομέα, αν και τα 21 δις τα οποία δόθηκαν και εκτός του τομέα αυτού δεν είναι και λίγα χρήματα, δεν έχουμε βγει ακόμα από την κρίση, γι' αυτό θα πρέπει σταδιακά να φύγουμε, αλλά όχι να διακόψουμε πλήρως όλα τα έκτακτα μέτρα και προγράμματα τα οποία είχαν ληφθεί. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου. Εμείς όταν δίνουμε την άδεια για ένα πρόγραμμα, έχουμε αξιολογήσει τους κινδύνους τους οποίους παρουσιάζουν αυτές οι τεράστιες προσπάθειες, Προσπαθήσαμε να δούμε να μην στηρίξουμε μία ανταγωνιστικού τομεί της οικονομίας αλλά και να αποτρέψουμε μία θα έλεγα πολυδιάσπαση της εσωτερικής μας αγοράς και να διασφαλίσουμε τη μη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Κάνοντας τα όλα αυτά θα βοηθήσουμε και την αύξηση του δυναμισμού μας του οικονομικού, την ανταγωνιστικότητά μας και να βελτιώσουμε τα δύσκολα δημοσιονομικά που αντιμετωπίζουν πολλές χώρες. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Προχωρώ κατευθείαν στον Επίτροπο Μπαρνιέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ε, ε, καλημέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε για την πρόσκληση ε, που μας κάνατε σε μένα και τον φίλο και συνάδελφο Αλμούνια και κάνοντας τις σωστές ερωτήσεις την κατάλληλη στιγμή θα προσπαθήσουμε να σας απαντήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και καταρχήν μιλάω για καλές ερωτήσεις γιατί πρέπει να δούμε ε, τι συνέβη κατά τα τελευταία δύο χρόνια και οι αναλύσεις οι οποίες ε, κάνατε κατά τον τελευταίο καιρό με τους συναδέλφους σας ε, η κυρία Πρόεδρε είναι ουσιαστικές και είναι η κατάλληλη στιγμή διότι υπάρχουν ορισμένες παράδοξες καταστάσεις αυτή τη στιγμή από τη μία πλευρά business as usual, σαν να μην τρέχει τίποτα και από την άλλη πλευρά για το θέμα που έθιξε ο Γιωακίμ, ε, για την ε, ε, συνέχιση των προβλημάτων. Θα ήθελα λοιπόν να αναφέρω τρία σημεία. Καταρχήν, ποια είναι η κατάσταση αγορά σήμερα. Δεύτερον, κατά τι τα μέτρα τα οποία λήφθησαν τελευταίως απέδωσαν. Και τρίτον, τι πρέπει να κάνουμε τώρα, τι έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε για να προλάβουμε μία ε, άλλη σημαντική δαπανηρή παρέμβαση, μαζική παρέμβαση των κρατών μελών. Φέρθηκε ο Χακίμ στις ε, κρατικές ενισχύσεις και δεν θα επανέλθω, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε πλέον να μιλάμε για την κρίση αυτή σαν κάτι παρελθόν, διότι ε, βέβαια βλέπουμε κάποια ανάπτυξη, ορισμένες αγορές που επανέρχονται σε φυσιολογική λειτουργία, ε, ορισμένες περιοχές έχουν σημαντικά κέρδη, δηλαδή φαίνεται ότι περάσαμε τη δύσκολη φάση και αυτό ήθελα να ε, πω και προηγουμένως αλλά είμαι ρεαλιστής και ως εκ τούτου ο πιο προσεκτικός γιατί διαπιστώνω τη μεγάλη αστάθεια των αγορών και ε, τις ε, διακοιμάνσεις των ε, πρώτων υλών δηλαδή θεωρώ ότι υπάρχει σημαντική κερδοσκοπία στις γεωργικές πρώτες ύλες υπάρχει ακόμη κάποια ανάρρωση του ευρώ πρέπει να δούμε τα μέτρα που λαμβάνονται στην Ιρλανδία και τέλος όπως και εγώ γνωρίζετε ότι υπάρχουν καταστάσεις και κοινωνικές οικονομικές επιπτώσεις ε, ε, που εκφράζονται στη μείωση ε, κατά τρεις μονάδες της αυξήσεως της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Οπότε η κατάσταση είναι ακόμη πολύ ευάλωτη και πρέπει να τελειώσει η έλλειψη διαφάνειας, η κακή αξιολόγηση των κινδύνων, να υπάρχει σταθερή λήψη ευθυνών για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αισιόδοξα το μέλλον. Στο δεύτερον, θα ήθελα να πω μετά το ε, Χοακίμ στο σημείο αυτό ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει λάβει τα έκτακτα απαραίτητα μέτρα για να μπορέσει να συμβάλλει στη δημιουργία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενός κλίματος ε, και ε, βλέπετε και εσείς όταν είσαστε υποψήφοι ε, στο γεγονός όπως είπα ότι η Ευρώπη κατάφερε να προστατεύσει τους πολίτες από την κρίση και καλύτερα ήταν να ήμασταν ενωμένοι για να λάβουμε τα μέτρα εκτός ε, και όχι ο καθένας για λογαριασμό του μόνος του. Κατά αυτόν τον τρόπο αποφύγαμε μία συστηματική κρίση ε, του ευρωπαϊκού συστήματος και ακόμη και αν στο παρελθόν πριν από την κρίση τα κράτη είχαν μπορέσει να εμποδίσουν την ανάληψη ε, ε, υπερβολικών κινδύνων όπως είδαμε στην αγορά των ακινήτων στην Αμερική. Από την άλλη πλευρά οι επόπτες δεν μπόρεσαν να εμποδίσουν τη συσσόρευση των κινδύνων που ε, απεκάλυψε η κρίση. Χρειάζεται λοιπόν να δούμε τις σωστές απαντήσεις και να αποφύγουμε το το ε, γεγονός ε, της μεταδόσεως ε, της ασθενείας και γι' αυτό πρέπει να αποδείξουμε στους Ευρωπαίους ότι η Ευρώπη προλαμβάνει και όχι μόνο θεραπεύει μία κρίση και να αποφύγουμε στο μέλλον τέτοιες καταστάσεις και το λέω αυτό διότι όλοι γνωρίζουμε ότι η δημοσιονομική μας κατάσταση δεν μπορεί να ανοιχθεί μία δεύτερη τέτοια κρίση και δεν θα το δεχθεί ούτε καν η δημόσια γνώμη και το κοινό. Γι' αυτό και μία ουσιαστική βαθιά αναθεώρηση του οικονομικού συστήματος θα μας επιτρέψει να προχωρήσουμε και γι' αυτό το επαναλαμβάνω όπως το είπα και στις 13 Ιανουαρίου δεν υποτίθεται ότι θα αναθεωρήσουμε διότι η κρίση ε, δεν ήταν ε, μία, ε, κάτι το υποτιθέμενο αλλά το, πραγματικά, το πραγματικό και γι' αυτό πρέπει να είστε βέβαιοι ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται πολύ αποφασισμένα για να αποφύγει να ξαναβρεθεί η Ευρώπη σε αυτή την κατάσταση. Δεύτερον, το θέμα της εποπτείας στην Ευρώπη για πιο αποτελεσματική εποπτεία. Και θέλω να σας πω ότι στο πακέτο της εποπτείας ο ρόλος σας ήταν αποφασιστικών για να δημιουργηθεί ένα ραντάρ για τους συστημικούς κινδύνους και να αποφύγουμε ε, ε, την κατάρρευση των των ε, εθνικών χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων. Ε, θα πρέπει βέβαια η Ευρώπη άπαξ και διατύπωσε τα μέτρα να τα χρησιμοποιήσει για να λειτουργήσουν. Ιδίω σε περίπτωση εντάσεων στην αγορά όπως το προτίμαμε με τον κανονισμό για το short selling. Και πάλι πρέπει να σας πω δημόσια ε, ότι το άρθρο 6 ε, του ε, κανονισμού ΕΣΜΑ θα ασχοληθεί με το θέμα αυτό. Η εποπτεία αναφέρεται και σε δύο πτυχές που θέλω να τονίσω. Καλύτερη εποπτεία των τραπεζών και ιδίως των μεγάλων τραπεζών και δεύτερον μία ανάλυση των συστημικών κινδύνων όπου πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να διασφαλίσουμε ότι οι συστάσεις της αρμοδίας επιτροπής θα εφαρμοστούν και δεν θα γνωηθούν. Είπα στον Υπουργό Οικονομικών προχθές στο Συμβούλιο ΕΚΟΦΗΝ ότι η Αμερικανική Επιτροπή των Συστηματικών Κινδύνων ε, συνήλθε για πρώτη φορά στην Αμερική ε, την περασμένη εβδομάδα. Δηλαδή είμαστε ε, στο ίδιο μήκος κύματος σε αυτό το σημείο. Και αυτή η εποπτεία είναι απαραίτητη αλλά δεν αρκεί για να μπορέσει το οικονομικό σύστημα να είναι υγιές. Πρέπει να το πράξουμε αλλά δεν αρκεί το μέτρο αυτό. Δεύτερον πρέπει να υπάρχει σωστή κεφαλαιοποίηση και αυτός είναι ο δεύτερος όρος τον οποίο προχωράμε μετά τη συμφωνία της Βασιλείας 3 για τους ίδιους πόρους και πηγαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα σας προτείνουμε την προσαρμογή αυτής της συμφωνίας ε, στις ε, αρχές του επομένου έτους. Θα το συζητήσουμε και αύριο το βράδυ σχετικά με την έκθεση του Ότμαρ Κάρα στην Ολομέλεια ε, και θέλω να χαιρετήσω την σημασία του. Η Συμφωνία της Βασιλείας αποτελεί ένα βασικό βήμα το οποίο όμως δεν πρέπει να βαρύνει υπερβολικά την οικονομία οικονομία και το σύστημα. Επιβεβαιώνουμε στο σημείο αυτό τις ε, μελέτες που έχουν γίνει για τις επιπτώσεις μικροοικονομικές και μακροοικονομικές για να μπορέσουμε να λάβουμε υπόψη μας τις ευρωπαϊκές ιδιομορφίες που πρέπει να προσαρμοστούν. Τρίτο βήμα είναι συχνά stress test, δηλαδή δοκιμασίες αντοχής για, τον, για τις τράπεζες και για τους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς διότι έγινε αυτό, ε, αυτή η πρώτη, ε, αυτός ο πρώτος γύρος των stress test για τις ε, τράπεζες είναι καλό εργαλείο το αποτέλεσμα φέτος το καλοκαίρι ήταν αποτελεσματικό και έγινε ε, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τους Ευρωπαίους επόπτες αλλά θα πρέπει να επαναλάβουμε την άσκηση αυτή. Τέλος, ε, τα εργαλεία για τη διαχείριση της κρίσεως, δηλαδή να μπορούμε για κάθε οργανισμό να έχουμε τα κατάλληλα ε, εργαλεία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα Οκτωβρίου θα παρουσιάσει μία συνολική ανακοίνωση και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω από αυτήν ορισμένες αρχές και θα δείτε ότι αντικατοπτρίζονται σε αυτή την ανακοίνωση. Καταρχήν, ότι όπως είπε η Λίζα Φερέρα, θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα διαχειρίσεως των κρίσεων σωστά. Δεύτερον, να έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να μπορούμε να επέμβουμε και ε, εγκαίρως να εντοπίσουμε τις τράπεζες οι οποίες μειονεκτούν προτού να χρειαστεί να τις σώσουμε και πολλά ε, μέτρα ε, βαίνουν προς αυτή την κατεύθυνση. Τρίτον να υπάρχει μία σαφής παρέμβαση σωστά οριοθετημένη. Τέταρτο εργαλείο θα, είναι, θα πρέπει ε, και οι πιστωτές και ε, οι μέτοχοι να συμβάλλουν τη στιγμή που θα χρειαστεί στα προγράμματα διασώσεως, δηλαδή θα πρέπει και οι τράπεζες να συμβάλλουν και θα δείτε σε αυτή την ανακοίνωση τα πρώτα εργαλεία για την συμβολή των τραπεζών κατά τρόπον ως το φορολογούμενος να μην είναι πάντοτε εις ε, την πρώτη γραμμή και να μπορούμε να επεμβαίνουμε σωστά για να μπορέσουμε σωστά να διαχειριστούμε την κρίση των τραπεζών που εκδηλώνονται συγχρόνως σε πολλά κράτη-μέλη, ξέρετε ότι πολλές από αυτές τις τράπεζες ανοίγουν σε κάποιο οργανισμό, όμιλο κάποια άλλης χώρας. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει η σωστή κατανομή των εξόδων και τέλος τα δικαιώματα του καθενός θα πρέπει να είναι καλά καθορισμένα εκ προημίου. Αυτά είχα να πω για την διαχείριση της, και αντιμετώπιση των κρίσεων των τραπεζών και προχωρούμε. Ακόμη και αν ακόμη δεν υπάρχει ομοφωνία, προχωράμε πολύ επικονομητικά στο Συμβούλιο των Υπουργών Οικονομικών. Καταλήγοντας λοιπόν πρέπει να σας πω ότι η πολύ σημαντική εργασία που έκανε ο συνάδελφος Αλμούνια επέτρεψε μαζί με τους συναδέλφους του Κοινοβουλίου να αποφύγουμε κρίσεις, ε, να αποφύγουμε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, να μπορέσουν οι τράπεζες να ε, αναδιαρθρωθούν εκ βάθρων και ελπίζουμε ότι όλα θα γίνουν με το σωστό ρυθμό και το ε, μάθημα που θα πρέπει να αποκονίσουμε είναι ότι πρέπει να αποφύγουμε να βαρύνουμε τους φορολογουμένους και να προλαμβάνουμε. Η πρόληψη κοστίζει πολύ λιγότερο από τη θεραπεία. Ως εκ τούτου πρέπει να είμαστε είμαστε σαφείς όσον αφορά την αγωγή και ε, τα φάρμακα για να αντιμετωπίσουμε και να στηρίξουμε τις τράπεζες οι οποίες κλειδονίζονται. Έχουμε μία αγορά όπου όχι μόνο οι τράπεζες δεν ε, χρειάζονται ε, το κράτος αλλά θα πρέπει να μπορούν να βοηθήσουν αυτούς οι οποίοι χρήζουν βοηθείας. Αυτό είναι η κατάληξή μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ περάσουμε τώρα στη συζήτηση. Είναι γεγονό ότι έχουμε καθυστερήσει λιγάκι και έχω ήδη μεγάλο κατάλογο μιλητών. Θα σας πω, έχω τον κύριο Μακάου, Φίλιπ Λαμπέτ, Μπουργκέζιο, Ίνετβελτ, Γκούλατ, Σάντσες Πρεσέντο, Τρεμόσα και Φόλφ Κλίντς. Αν θέλει κανείς άλλος να πάρει το λόγο και το ξέχασα, παρακαλώ να μου το πει. Κλείνω τότε τον κατάλογο των ομιλητών. Ο κύριος Σιμών επίσης. Κλείνω τον κατάλογο των ομιλητών. Παρακαλώ να είστε σύντομοι, ένα λεπτό για κάθε ερώτηση και παρακαλώ να πείτε σε ποιον επίτροπο απευθύνεστε. Σε ομάδες τριών θα ακούσουμε τις ερωτήσεις και μετά θα περάσουμε σε απαντήσεις. Ποιος είναι πρώτος. Ευχαριστώ πολύ. Σεβαστήκαμε την εσωτερική αγορά προκειμένου να μην υπάρχει στρέβλωση του ανταγωνισμού. Δεν μας είπε ο Επίτροπος πώς ακριβώς όμως έγιναν τα πράγματα. Δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα των τραπεζών που είναι σημαντικά, αλλά πρέπει να δούμε και πώς φτάνουν οι πιστώσεις στις οικογένειες και στις εταιρείες. Και αν δεν συμβαίνει αυτό, για ποιο λόγο και για, για την αναδιάρθρωση. Ο Επίτροπος Αλμούνια μας λέει ότι θα παραταθεί το προσωρινό πλαίσιο με κάποιους επιπλέον κανόνες. Τι δεν λειτουργήσε όμως, τι ακριβώς πρέπει να τροποποιηθεί και για ποιο λόγο. Μία ερώτηση προς τους δύο επιτρόπους. Συνεργάζεστε σε σχέση με αυτό το προσωρινό πλαίσιο λοιπόν αναδιάρθρωσης, ε, η συνεργασία σας θα συνεχιστεί ή έχετε και ξεχωριστό πρόγραμμα ο καθένας. υπάρχει και το θέμα της εποπτείας. Στην αρχή μιλήσαμε για μια ανακοίνωση για τον Οκτώβριο και μάλιστα είχαμε πει ότι θα ισχύσει από τώρα, από το φθινόπωρο. Μου φαίνεται ότι έχουμε λίγο καθυστερήσει. Είδαμε τι έγινε και στην Ιρλανδία. Πότε πιστεύετε ότι θα μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση και συνεπώς από τα προσωρινά αυτά μέτρα. Πότε θα έχουμε ολοκληρωθεί, ολοκληρώσει με την ε, ε κακή κατάσταση της οικονομίας. Προς τον κύριο Αλμόνια, ο κύριος Λαμπέρτς. Μιλήσατε για τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ε, για τις ε, κρατικές ενισχύσεις. Ε, πολλές φορές μας ρώτησαν σε ποιο βαθμό, κατά την άποψή σας, τα μέτρα που ελήφθησαν από την ΕΚΤ μπορούν, συνιστούν στρέβλωση του ανταγωνισμού. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Οι υπηρεσίε σα και απευθύνομαι και στον κύριο Μπαρνιέ έχουν κάνει μια αξιολόγηση του τι θα σήμαινε in fine το καθαρό κόστο για τα κράτη-μέλη. Ενδεχομένω να είναι πολύ νωρί να το πούμε αυτό. εσεί. λέτε όμω ότι όλα αυτά δεν επικερδεί για τα κράτη-μέλη τελικά ε, κάνατε μια αξιολόγηση να δείτε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση και αν τελικά οι καθαρές εισρωές ε, έχουν όντως φτάσει στις τράπεζες ή όχι. Επίσης αναφερθήκατε στα τεστ αντοχής. Η Allied Irish Bank, έμαθα, η οποία σιγά σιγά ε, καταραίει, πέρασε το τεστ αντοχή όμω. Και θα ήθελα να μου πείτε ποια είναι η δική σα ανάλυση, γιατί τι νόημα έχει να έχουμε τεστ αντοχή, αν μετά τελικά διαπιστώνουμε ότι δεν εξυπηρετούν σε τίποτα. Και επίση για τη Βασιλεία 3, Εμάς μας ανησυχεί η περίοδος ε, η μεταβατική και θα ήθελα να μου πείτε αν συμφωνείτε με το γεγονός ότι ανεξαρτήτως από τη ε, διάρκεια της περίοδου μετάβασης ε, να, μην, να, ισχύσουν σοβαρές, ε, σοβαροί όροι για τις τράπεζες οι οποίες ε, δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Κοιτάξτε, δεν είναι ανταγωνισμός για το πόσε ερωτήσεις θα χωρέσετε σε μία ερώτηση, γιατί, σε ένα λεπτό, γιατί τελικά δεν θα μπορέσετε να πάρετε τις απαντήσεις. Θα ήθελα να σας πω λοιπόν ε, να είστε πιο σύντομοι. Ο κύριος Ευχαριστώ. Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Στα πλαίσια των πολλαπλών λύσεων για να πάψουν να είναι υπερχρεωμένα τα κράτη, Ο καθηγητής Αρτούς της Νατεξής έχει προτείνει μια ενδιαφέρουσα λύση. Ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του χρέους να περάσει στην κεντρική τράπεζα που στην ουσία ε, θα ε, παρουσιάσει με διαφορετική μορφή το δημόσιο χρέος. Οπότε μήπως έτσι θα μπορούσαμε να ακυρώσουμε ένα κομμάτι του δημοσίου χρέους. Αυτό βέβαια θα επιβαρύνει τον ε, προϋπολογισμό της Κεντρικής Τράπεζας αλλά θα ελαφρύνει ουσιαστικά τους Ευρωπαίους αποταμιευτές και πολίτες. Εμείς ζητάμε επίσης σαν Ευρωπαϊκή Ένωση να υπάρξει ανατίμηση του Ιουάν. Ε, τι ακριβώς γίνεται εδώ. Νομίζω ότι έχετε αποφασίσει, έχετε συζητήσει κάποιες ενέργειες για να αντιμετωπιστεί αυτή η επιθετική και μη ανταγωνιστική πολιτική που προέρχεται όχι μόνο από την Κίνα αλλά και από τις Ηνωμένε Πολιτείες. Κύριε Αλμούνια, θα είστε ο πρώτος που θα δώσετε απαντήσεις. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο σύντομος όσο και αυτοί που έβαλαν πέντε ερωτήσεις σε λιγότερο από ένα λεπτό. Για τον κύριο Μαργκάγιο, είναι σαφές ότι σεβόμεθα τις βασικές αρχές οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν. Βέβαια υπάρχουν σοβαρότατα προβλήματα στον χρηματοπιστωτικό τομέα Ξέρετε ότι από την αρχή της κρίσης τα πράγματα είναι δύσκολα. Παρ' όλα αυτά σεβαστήκαμε τις αρχές αυτές. Προφανώς λάθη έχουν γίνει. Άνθρωποι είμαστε, αν και επίτροποι που κάνουμε λάθη. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν είχε αναλάβει δράση όταν συζητούσαμε τα εθνικά προγράμματα και τις μεμονωμένες περιπτώσεις, τότε σήμερα τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ άσχημα, θα είχαμε μια εσωτερική αγορά στα πλαίσια της οποίας η χρηματοπιστωτική γενικά δραστηριότητα θα είχε ακυρωθεί. Τα κράτη-μέλη έχουν πάρει φυσικά και κάποια μέτρα με πάρα πολύ ψηλά ποσά και έχουν αναλάβει συγκεκριμένους κινδύνους να διατρέξουν στο όνομα των φορολογουμένων πολιτών κάθε φορά. Όμως αν δεν είχε γίνει κάτι τέτοιο θα είχαμε πράγματι μια τεράστια στρέβλωση στον τομέα και κάποιες τράπεζες οι οποίες θα κατέστρεφαν ουσιαστικά με τις συμπεριφορές τους στην αγορά. Παρ' όλα αυτά αυτοί οι κίνδυνοι δεν έγιναν πραγματικότητα και χάρη στις ε, ενέργειες τις δικές μας. Μιλήσατε και για τις ροές των πιστώσεων. Υπάρχουν ορισμένοι αριθμοί που δείχνουν μια κάποια τάση προς ανάκτηση μιας κάποιας ταχύτητας. Αλλά για να λειτουργήσει το σύστημα σωστά από εδώ και πέρα χρειαζόμαστε ισχυρές τράπεζες και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε κάπως υπομονετικοί. Υπάρχουν κίνδυνοι ακόμα και δεν έχει εξομαλυνθεί πλήρως η κατάσταση όταν τίθενται τα ερωτηματικά αυτά προς τους τραπεζίτες, ε, μας λένε ότι τελικά μας ζητούν πιστώσεις οι οποίες ε, δεν μπορούν να δοθούν, δεν μπορούμε να δανείσουμε αυτούς που θέλουν να τους δανείσουμε γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα να μας τα επιστρέψουν. Ενώ εμείς θα θέλαμε να δανείσουμε κάποιους άλλους που έχουν αυτή τη δυνατότητα αλλά δεν μας ζητούν να τους δανείσουμε. Λοιπόν, σας είπα ότι ε, θα υπάρξουν κάποιες ε, διακοπές των δυνατοτήτων οι οποίες υπήρχαν μέχρι τώρα, μέχρι το ποσό των 500.000 ευρώ σχετικά με τις κρατικές βοήθειες. Αυτό το κατώτατο όριο ε, δεν θα συνεχιστεί να ισχύει. Βέβαια όταν πρόκειται για κάποιες εγγυήσει ίσως τα πράγματα να συνεχίσουν να ισχύουν και του χρόνου. Θα δείτε ότι οι διαφορές καταρχάς στα επιτόκια ανάμεσα στις διάφορες χώρες δεν είναι πάρα πολύ μεγάλες. Η κατάσταση δεν έχει εξομαλυνθεί πλήρως. Ε, θα δούμε τι θα γίνει επίσης και με τα λεγόμενα πράσινα προϊόντα γιατί δεν έχουμε χρησιμοποιήσει τις δυνατότητες τις οποίες είχαμε μέχρι εκεί. Δεν έχει υπάρξει και αντίστοιχη, θα έλεγα, χρήση των δυνατοτήτων που είχαμε σε σχέση με τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε ε, να ορίσουμε το πλαίσιο, το προσωρινό και για το 2011 σχετικά με τις μικρομεσαίες. Το πλαίσιο που ισχύει μέχρι σήμερα θα δούμε αν θα ισχύσει και του χρόνου συνεργαζόμεθα και με τον Επίτροπο Μπαρνιέ και με τις άλλες υπηρεσίες και γενικές διευθύνσεις. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στη συνεργασία μας. Υπάρχει μεγάλη βούληση συνεργασίας και το ίδιο ισχύει και με τον Επίτροπο Όλη Ρένα και την διεύθυνση στην οποία προείσταται, την οποία γνωρίζω καλά λόγω των παλαιών μου αρμοδιοτήτων. Λοιπόν, βγήκαμε από την ύφεση, θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά δεν βγήκαμε ακόμα από την κρίση. Οι συνθήκες είναι δύσκολες. Για τον κύριο Λάμπερτς τώρα. Νομίζω ότι η νομισματική πολιτική δεν είναι κρατική βοήθεια. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η κρατική βοήθεια από τη μία και η νομισματική πολιτική από την άλλη. Αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρχίσει να ανακατεύεται στα νομισματικά θέματα, ε, τότε έχει τελειώσει πλέον η ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας. Θα πρέπει λοιπόν μετά από αυτή την κρίση να κάνουμε μια αξιολόγηση του τρόπου με τον οποίο ασκεί την νομισματική πολιτική η Κεντρική Τράπεζα. Τα θέματα αυτά άπτονται της πολιτικής της νομισματικής όπως επίσης και της ανεξαρτησίας της Κεντρικής Τράπεζας το κόστος της κρίσης, το συνολικό. Είναι νωρίς ακόμα για να καταλήξουμε σε ένα αριθμό. Θα δούμε αν ας πούμε οι εγγυήσει οι οποίες έχουν δοθεί θα χρησιμοποιηθούν και σε ποιο μέτρο θα χρησιμοποιηθούν. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα τελικό ποσό. Έχουν υπάρξει ενέσεις δημοσίου κεφαλαίου, τις οποίες κάποια στιγμή ελπίζουμε να επιστραφούν. Θα δούμε τώρα με ε, πώς τα κράτη-μέλη θα αντιμετωπίσουν αυτή την εκ νέου διάθεση των κονδυλίων. Είναι εν πάση περιπτώσει νωρί για να μιλήσει κανείς για το τελικό κόστος της κρίσης. Γνωρίζουμε όμως τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα χρήματα του δημοσίου, των πολιτών, των φορολογουμένων που χρησιμοποιούνται στην αντιμετώπιση της πιστοτικής κρίσης. Όπως σας είπα στους αριθμούς που ανέφερα προηγουμένως μιλάμε για πάρα πολύ χρήμα αλλά ναι μεν πολύ χρήμα, αλλά είναι δύσκολο να πούμε τι θα χάσουμε και τι θα κερδίσουμε στο τέλος, όταν γίνει ο τελικός λογαριασμός. Στη δεκαετία του 90 είχαμε κάποια παραδείγματα όπου παρεμβάσεις τέτοιες κρατικές κέρδισαν τελικά. Το κράτος διακινδύνευσε αν θέλετε τα χρήματα των φορολογουμένων αλλά βγήκε σε καλό αυτό. Μιλήσατε για την Irish Bank. Δεν κινδυνεύει έτσι η τράπεζα αυτή. Είναι μια τράπεζα που ε, ε, που λύνει τα προβλήματά της. Το πρόβλημα στην Ιρλανδία είναι η Anglo-Irish αν ακούσαμε καλά και όχι η Allied Irish. Τώρα σχετικά με το δημόσιο χρέος πώς μπορούμε να το στείλουμε όλα στο, στην κεντρική τράπεζα αυτή είναι μια ψευδολύση, δεν θα λύσει τίποτα. Περί, περίμενε να απαντήσω Κοιτάξτε, διακόπτει ο κύριος Μποργέζιο. Εγώ είπα ένα τμήμα του δημοσίου χρέους να πάει στην Κεντρική Τράπεζα. Κοιτάξτε, αυτό το οποίο κάνει η Κεντρική Τράπεζα είναι να αγοράζει τίτλους που έχουν σχέση φυσικά με το δημόσιο χρέος τη ζώνη ευρώ ανάλογα με το τι απαιτούν οι συνθήκες. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε ε, αυτή τη στιγμή αγοράζουν επίσης και ε, κρατική δημόσια παρέμβαση της Ελλάδας, της Πορτογαλίας και της Ιρλανδίας. Εν πάση περιπτώσει αυτά τα αποφασίζει η Κεντρική Τράπεζα και εσείς όταν έχετε τον κύριο Τρισέ εδώ θα τον ρωτάτε τι κάνει και πόσο και για πόσο καιρό σχετικά με τις ισοτιμίες. Νομίζω ότι σήμερα η Τρόικα, ο Γιούνκερ, Ρεν και Τρισέ συζητούν ακριβώς τα θέματα αυτά Ελπίζω να είναι χρήσιμη η συνάντηση που θα έχουν με τον Πρωθυπουργό της Κίνας. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχήν να σας πω ότι αντιλαμβάνουμε την ανυπομονησία σχετικά με την ε, πρόταση της Επιτροπής ε, σχετικά με την διαχείριση και την πρόληψη των κρίσεων αλλά τα πράγματα θα προχωρήσουν όπως σας είπα σοβαρά, γρήγορα, καλά και χωρίς να αυτοσχεδιάζουμε. Θα κάναμε ένα πρώτο σχέδιο, θα το συζητήσουμε γύρω στις 20 Οκτωβρίου θα κάνουμε μία δεύτερη ανακοίνωση και είχα δύο ε, δυνατότητε να συζητήσω με τους ε, αρμόδιους υπουργούς τελευταία στη Μαδρίτη και την Άνοιξη θα παρουσιάσουμε τις νομοθετικές προτάσεις. Γιατί κύριε Γκαρσία Μαργκάλιο πρέπει ε, να πάρουμε αρκετό χρόνο, γιατί είναι περίπλοκο το θέμα, είναι τα δικαιώματα των πιστωτών. αν κοιτάξουμε ε, τα 27 συστήματα χρεοκοπίας ε, ή στην Ευρώπη και να προσπαθήσουμε να τα εναρμονίσουμε. Δεν μπορούμε να αυτοσχεδιάζουμε. Ο χρόνος λοιπόν τον οποίο ε, θα αφιερώσουμε όπως έγινε και με τα χρηματοοικονομικά παράγωγα και με άλλες περιπτώσεις να είστε βέβαιος ότι το καλοκαίρι εποφελήθηκα για να δουλέψω και να παρουσιάσω κείμενα τα οποία εις αντίθεση με τους Αμερικανούς να μπορέσουν ε, να ισχύσουν και να βοηθήσουν την εργασία σας. Λοιπόν, ε, ήθελα να σας πω ότι θα υποφεληθώ για να σας παρουσιάσω το πιο πλήρες δυνατό κείμενο. Κύριε ε, Λαμπέρ, όπως ξέρετε η Anglo-Irish δεν είχε εξεταστεί γιατί ήταν εθνικοποιημένη. Η Allied Irish πέρασε το τεστ όπως είπατε αλλά το stress test έγινε μια δεδομένη μέρα. Δεν ε, ισχύει για πάντα. Γι' αυτό σας είπα και προηγουμένως ότι θα πρέπει να προσιλωθούμε και να επαναλαμβάνουμε αυτές ε, τις ε, δοκιμασίες για να δούμε και να συγκρίνουμε με την προηγούμενη περίοδο για να υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια. Διαπιστώνω ότι ε, μία ε, προς μία οι τράπεζες ε, και οι αρχικές αρχές αναλαμβάνουν μέτρα αναδιαρθρώσεως όπως έγινε και στην Ιρλανδία. Για τη δεύτερη ερώτησή σας η απάντησή μου είναι θετική. Ναι. Αυτό ακριβώς με απασχολεί, αυτό ετοιμάζω χωρίς να αυτοσχεδιάζω κατά τρόπον ώστε στο, στην εργαλειοθήκη αυτή να μπορέσουμε να υποφεληθούμε από όλα τα συμπεράσματα των ερευνών μας για να έχουμε τα σωστά εργαλεία στην εργαλειοθήκη. Δηλαδή όταν διαπιστώνεται ένας κίνδυνος ή μία άτυπη συμπεριφορά θα υπάρξει απαγόρευση ορισμένων τραπεζικών των ε, ε, λειτουργιών, θα αλλάξει η διαχείριση, ε, θα ζητηθεί να συμβάλλουν οι μέτοχοι, οι πιστωτές και θα πρέπει να διαρθρώσουμε το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινούμαστε. Βλέπετε λοιπόν ότι υπάρχουν σοβαρές προϋποθέσεις στην εργαλειοθήκη αυτή την οποία θα σας παρουσιάσω μέσα Οκτωβρίου. Θα ήθελα επίσης να προσθέσω κάτι σε αυτά τα οποία πολύ σωστά υπόχω ο Αλμούνια Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο θεωρούμε ως πάρα πολύ σοβαρό. Είναι το ε, οικονομικό σύστημα και η αστάθειά του. Ο κύριος Γιούνκερ και ο κύριος Τρισέ σήμερα συναντούνται με τις ε, κινέζικες αρχές και ε, επιζητούμε ένα πιο ακριβές σύστημα κατά τρόπον ώστε να μπορέσει κανείς να έχει μέτρα για το μέλλον ε, διότι όπως ξέρετε ότι η Κίνα έχει λάβει τα πρώτα μέτρα που είναι στη σωστή κατεύθυνση και δεδομένου του ρόλου που θα παίξει στο πολιτικό και διπλωματικό χώρο ε, και εφόσον είναι ένας από τους παγκόσμιους πρωταγωνιστές θα πρέπει να την ενθαρρύνουμε να λαμβάνει τα σωστά μέτρα προς τη σωστή κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Επόμενος γύρος ερωτήσεων, ε, η Σόφη, η Σιλβή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πέρσι, όταν ε, εγκρίναμε την έκθεση, την έκθεση την ετήσια έκθεση ανταγωνισμού 2008 ζητήσαμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας κάνει μια περιστατωμένη ανάλυση του αντικτύπου των κρατικών ενισχύσεων. Και κάθε φορά έχουμε απλώς μια σύνοψη των, αποφάσεων που έχουν ληφθεί, αλλά δεν μαθαίνουμε τίποτα για τα αποτελέσματα. Καταλαβαίνω ότι είναι σύντομα, αλλά, αλλά εάν ξοδεύουμε τόσο πολλά δημόσια χρήματα, είναι χρήσιμο να ξέρουμε κατά πόσο ξοδεύονται σωστά. Μήπω την παρουσίαση δεν το πήρα είδηση, αλλά βλέπω και πάλι τις σημειώσεις ε, και βλέπω και πάλι μια λίστα με, αποφασ... με αποφάσεις. Έχουν δοθεί τόσα χρήματα στο ένα ή στο άλλο πρόγραμμα, αλλά δεν ξέρω αν έχουν σωστά δαπανηθεί τα χρήματα αυτά. Και μόνο αν κάνουμε την ανάλυση αυτή μπορούμε να δικαιολογήσουμε ε, την εισαγωγή, την κατάργηση ε, μέτρων, την τροποποίηση των μέτρων. Δεν κατάλαβα πολύ καλά εάν τελικά τροποποιήσατε ή αν περιορίσατε ακόμη περισσότερο το, περισσότερο το, προσωπικό, το προσωρινό πλαίσιο. Εμάς το Κοινοβούλιο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό, γιατί μιλάμε για ποσά τεράστια που έχουν ε, αυξήσει, έχουν διωγγώσει το δημόσιο χρέος και θέλουμε να ξέρουμε αν ήταν χρήσιμη η ε, δαπάνη των ε, ποσών αυτών. Ευχαριστώ πολύ. Ε, να συνεχίσω αυτά που είπε η Σοφή Ίνετφελτ. Ε, είμαστε σε μια έκτακτη περίπτωση, εξαιρετική περίπτωση. Δεν λέω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολύ καλώ έκανε ό,τι έκανε, αλλά όταν βρισκόμαστε στην εξαίρεση και όχι στον κανόνα και όταν, φτάμε για, όταν φτάνουμε σε τέτοια ποσά, ε, νομίζω ότι έχουμε το δικαίωμα να ξέρουμε πού πήγαν τα χρήματα αυτά και επίσης να μπορούμε να πούμε στους πολίτες μας τι τα κάναμε. Ενδεχομένως ο κύριος Μπαρνιέ να θέλει να μου απαντήσει σε αυτό. Αλλά σε μία κρίση πρέπει κάποιος να εξελιχθεί. Πρέπει, κάπου, πρέπει να προστατευτούμε. Ε, ε, θα πρέπει τα παιδιά μας να, θα πρέπει για τα παιδιά μας να προστατεύσουμε και το παρόν. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να υποθηκεύουμε χρήματα για κάτι που δεν υπάρχει. Καταλαβαίνω αυτό που είπατε, ότι εντάξει η ανάπτυξη μπορεί να μην ήταν ε, το βασικό μέλημα όσων πήραν τα χρήματα. Τι τα κάνουμε όμως αυτά τα χρήματα, τι κάνουμε, προστατεύουμε το παρελθόν σε έναν κόσμο που όλα αλλάζουν συνεχώς ή προσανατολισμό, προσανατολιζόμαστε σε μελλοντικές λύσεις. Καταλαβαίνω τη δυσκολία, ε, καταλαβαίνω ότι χειρίζεστε σε μια δύσκολη περίοδο την ευρωπαϊκή οικονομία, αλλά θέλουμε και ποιοτικό, ποιοτική, ε, ποιοτικό κατάλογο και όχι μόνο ποσοτικό όταν έρχεστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Χαίρομαι πολύ που είναι εδώ οι δύο επίτροποι. Είναι γεγονό ότι έχουμε προσωρινά μέτρα και συνεπώς πρέπει να έχουμε και μία ε, επίβλεψη των μέτρων αυτών. Είναι λοιπόν πολύ χρήσιμη η παρουσία των δύο επιτρόπων. Είναι γεγονό ότι είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία επίγουσα κατάσταση. Κάποια μέτρα παρουσιάζουν προβλήματα σήμερα, ενδεχομένως κάποια να επιδεινώνουν και την κρίση. Γι' αυτό πρέπει να προσπαθήσουμε να δούμε πώς μπορούμε να τα προσαρμόσουμε τα μέτρα αυτά σύν χρόνο. Μία ερώτηση όσον αφορά τη συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Θα ήθελα να μου πείτε για την αποδοτικότητα των μέτρων αυτών. Υπάρχουν κάποια προβλήματα οικονομικής φύσεως, γιατί μερικές φορές ε, μπορεί να καθυστερεί η προσαρμογή των μέτρων αυτών. Μιλήσαμε για ε, καλύτερη εφαρμογή, για πιο αυστηρή εφαρμογή των μέτρων. Ίσως θα έπρεπε να έχουμε περισσότερα μακροπρόθεσμα μέτρα. Ίσως θα μπορούσατε εσείς να μας πείτε περισσότερα από αυτού όσον αφορά τις ενισχύσεις και τη χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Συμφωνούμε απολύτω με την απόφαση αυτή, είναι πολύ σημαντικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Πρέπει και εκείνες να μπορούν να υποφεληθούν από κάποια μέτρα και όχι πάντοτε να περνούν από οικονομικούς ενδιάμεσους για να το επιτύχουν αυτό. Μιλήσατε κύριε Παρνιέ για το τι έγινε σε επίπεδο εποπτείας ε, και ρύθμισης. Τώρα αυτά όμως πρέπει να γίνουν πράξη. Από απόψεως χρονοδιαγράμματος, ποια είναι τα μελλοντικά μέτρα για να μην για να μην μείνουμε μόνο στα λόγια για να περάσουμε στην πράξη. Πρόεδρος, ο κύριος Μπαρνιέ, πρώτα το λόγο, ε, θα έχει πρώτα το λόγο, γιατί οι περισσότερες ερωτήσεις απευθύνθηκαν και γίνουν. Ίσως ε, ο Ζωακίμ να απαντήσει ε, με περισσότερες λεπτομέρειες σε κάποιες από τις ερωτήσεις, όπως αυτές που έθεσε η Σιλβί Γκουλάρ. Στα πλαίσια της προσπάθειας την οποία κάνουμε σήμερα βλέπετε ότι από τη μία ο κύριος Σαλμούνια στα πλαίσια των ευθυνών του εξηγεί το πόσο διαχειριστήκαμε στο πρόσφατο παρελθόν τις βοήθειες που δόθηκαν. Εγώ ε, που συνεργάζομαι μαζί του πιστεύω αρμονικά προσπαθώ μαζί σας να οικοδομήσουμε ένα σύστημα σύμφωνα με το οποίο δεν θα έχουμε ανάγκη από τέτοιου είδους βιοήθειες στο μέλλον. Αυτή είναι η προσπάθεια την οποία κάνουμε. Εμείς δεν θέλουμε να αρκεστούμε σε ρυθμίσεις, σε περιόδους κρίσης και σε εξυγίανση της οικονομικής διακυβέρνησης. Θέλουμε να μιλήσουμε απευθείας στον Ευρωπαίο πολίτη για ένα πρόγραμμα οικονομικό που να γεννά <coughs> απασχόληση, ανάπτυξη, έτσι ώστε η ανάπτυξη την οποία θα επιδιώξουμε να είναι πιο ποιοτική, να είναι πιο πράσινη από αυτήν τουλάχιστον που είχαμε τα τελευταία 15 χρόνια. Αυτή είναι η φιλοσοφία να συνεργαστούμε μαζί σας, έχετε ένα μείζωνα ρόλο να παίξετε και να οικοδομήσουμε νέους κανόνες. Και στην ουσία να ξαναφέρουμε τις χρηματαγορές στην πραγματική οικονομία και όχι το αντίθετο, γιατί αυτό βλέπουμε εδώ και 15 χρόνια. Οι χρηματαγορές θα πρέπει να ενταχθούν σε ε, μακροπρόθεσμες επενδύσεις, όχι να επιδιώκουμε συνέχεια το μέγιστο δυνατό κέρδος στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Αυτή είναι η στρατηγική την οποία θα ακολουθήσω τα επόμενα χρόνια. Να ξαναβάλουμε τις χρηματαγορές εκεί όπου δεν έπρεπε ποτέ, από όπου δεν έπρεπε ποτέ να βγούνε την πραγματική οικονομία. Θα πρέπει δηλαδή οι χρηματαγορές να εξυπηρετήσουν την πραγματική οικονομία στα πλαίσια φυσικά της ενιαίας αγοράς για την οποία έχουμε τη συλλογική ευθύνη. Θα σας παρουσιάσουμε και το λεγόμενο Single Market Act ξανά σε μερικούς μήνες. Θέλουμε η ενιαία αυτή αγορά να λειτουργήσει καλύτερα για μεγαλύτερες επενδύσεις, για ανάπτυξη, για ανανταγωνιστικότητα και κυρίως για την ποιοτική βελτίωση της ζωής των πολιτών, είτε είναι εργαζόμενοι, καταναλωτές, πολίτες, αποταμιευτές, χρήστες δημοσίων υπηρεσιών. Αυτός είναι ο στόχος μας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ένα δεύτερο τμήμα των ευθυνών, στα πλαίσια πάντα των συνεργασίας μου με τον Ιωακήμ και με άλλους συναδέλφους, είναι να οδηγηθούμε σε μια νέα μορφή ανάπτυξης. Θυμίζω προς την κυρία Γκουλαρό ότι για να μπορέσουμε αυτή, αυτή, αυτόν τον νέο διακανονισμό και αυτή τη νέα εποπτεία στην οποία καταλήξαμε, είναι στόχος μου να θέσω στη διάθεση αυτών που παίρνουν αποφάσεις τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις το ένα σύνολο προτάσεων, χρήσιμων ελπίζω, μέχρι την επόμενη άνοιξη. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και ο χρόνος που περνά, ε, παρότι έχουμε θα έλεγα σε εισαγωγικά μικρή μνήμη, κοντή μνήμη όλοι, πρέπει να ε, εκμεταλλευτούμε το χρονικό αυτό διάστημα και να μην ξεχάσουμε τίποτα από ό,τι έχουμε περάσει και κάνει μέχρι τώρα. Προσπαθούμε λοιπόν και σε τεχνικό επίπεδο και σε δημοσιονομικό επίπεδο οι τρεις αρχές ε, τις οποίες ε, βοηθήσατε να δημιουργηθούν να δουλέψουν από την 1η Ιανουαρίου. Τις πρώτες εβδομάδες θα λειτουργήσουν με διευθυντές οι οποίοι θα λειτουργήσουν με τη σειρά τους μεταβατικά και αυτό ισχύει και για το Συμβούλιο Συστημικών Κινδύνων ε, θα πρέπει να τα προετοιμάσουμε όλα αυτά και να ετοιμάσουμε και τον μικρό κατάλογο, το συνοπτικό κατάλογο, το short list των προσωπικότητων με δύο βασικά κριτήρια. Την ανεξαρτησία από τη μία και την επαϊωσύνη από την άλλη. Λοιπόν, αυτές είναι οι προτεραιότητες μου έτσι ώστε να κάνω πραγματικότητα αυτά τα οποία εσείς ψηφίσατε. Είστε έτοιμος? Ωραία. Λοιπόν, στην κυρία Ίνβελτ όσον αφορά την ε, επίπτωση της ε, κρατικής ενίσχυσης. Είναι πολύ νωρίς. Δεν έχουμε ε, εξέλθει ακόμη για να μπορέσουμε να κάνουμε απολογισμό του ό,τι κάναμε κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου. Νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς. Μπορούμε να έχουμε μία πρόχειρη αξιολόγηση για την οικονομική πτυχή αυτής της μεγάλης προσπαθίας. Αποφύγαμε ε, την καταστροφή μπορέσαμε να βοηθήσουμε και να αναδιαρθρώσουμε πολύ δύσκολες καταστάσεις στον οικονομικό τομέα με ορισμένα πιστοτικά ιδρύματα. Είδαμε ότι βρήκαμε με την ε, κρίση αυτή τι δεν υπήρχε, τι δεν προβλεπόταν στον, ε, στο πλαίσιό μας και με την συνεργασία σας όντως εντοπίσαμε τι χρειάζεται ακόμη και τι πρέπει να προχωρήσουμε στους επόμενους μήνες και χρόνια για να μπορέσουμε να είμαστε ασφαλείς. και να αποφύγουμε αυτόν τον ε, κίνδυνο. Αλλά είναι κάτι ε, το οποίο ε, έχει γίνει στο σύστημα, στον οικονομικό τομέα με το σύστημα που είχαμε, που ήταν οι κρατικές ενισχύσεις, που δεν είχαν προβλεφθεί καν για αυτές τις καταστάσεις. Οπότε επινοήσαμε το, ένα πλαίσιο για έκτακτες καταστάσεις που βασίζεται σε αυτή την έκτακτη νομική βάση προσπαθήσαμε να αποφύγουμε τους κινδύνους που επεσήμανα προηγουμένως και ακόμη διαχειριζόμαστε πολύ δύσκολα θέματα και προηγουμένως ε, μιλήσαμε για την Ιταλία για την Ιρλανδία με συγχωρείτε αλλά η Landesbank πόσα χρόνια ήταν η συνήθις ε, ύποπτη ε, για τους ε, επιτρόπους και τώρα ασχολούμεθα με τις οροφές, με τα προβλήματα αυτών των ο τραπεζών και χρησιμοποιούμε τα εργαλεία που έχουμε για να ε, επέμβουμε εις βάθος αυτές τις τράπεζες. Επίσης αποφασίσαμε και ε, συγκεκριμένα πράγματα σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Η Φόρτις παραδείγματο χάρη. Στην ε, κρίση της Φόρτις είδαμε ότι η μόνη λύση ήταν να υπάρξει κατακαιρματισμός στον πυρήνα της εσωτερικής αγοράς, στον Μπενελούξ, στους ιδρυτές της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τώρα παρακολουθούμε το, την εφαρμογή των μέτρων που αποφασίστηκαν και είναι ε, εύκολο να αποφασίσουμε διότι οι εθνικές αρχές συμμορφώνονται 100% με τις αποφάσεις που λαμβάνουμε αλλά σε άλλες καταστάσεις ξέρετε ότι αυτό δεν είναι εύκολο κάνουμε όμως ό,τι μας είναι δυνατόν και πιέζουμε όσο είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε ε, την εφαρμογή των αποφάσεων που πήραμε άλλη πλευρά της οικονομίας, στο προσωρινό πλαίσιο όπως είπα, με τη δικιά μας ανάλυση η οποία δεν μπορεί να είναι η τελική ε, για το πλαίσιο των ε, έξι κεφαλαίων. Εμείς είχαμε πει ότι μετά τις 31 ε, Δεκεμβρίου πρέπει να τελειώσουν οι 500.000 ευρώ βοήθεια να εταιρεία. Δεν είναι καλό, δεν πρέπει να προχωρήσει διότι όπως είπε και ο κύριος Γκαρσία Πρεσέντο θα παρατείνει την κατάσταση και ε, θα εμποδίσει τις αναγκαίες προσδιαρμογές. Δεν είναι χρήσιμο λοιπόν. Ήταν αναγκαίο ίσως ε, στην πιο δύσκολη στιγμή της κρίσεως. Τώρα όμως δεν χρειάζεται άρα θα τελειώσει. Επίσης με τις επιχορηγούμενες πιστώσεις ή εγγυήσεις ε, ε, ε, δεν μπορούσε κανείς να εφαρμόσει την κατευθυντήρια γραμμή για τις κρατικές ενισχύσεις. Οπότε με ορισμένες εξαιρέσεις αποφύγαμε τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτά τα μέτρα για μεγάλες εταιρείες που είχαν λιγότερα προβλήματα να έχουν πρόσβαση τις επιστώσεις και να τις επικεντρώσουν περισσότερο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα πρέπει υπό αναθεωρημένες συνθήκες πιο αυστηρές και για το 2011 να παράσχουμε κάποια βοήθεια διότι δεν θα έχουν ε, ατελείωτη πρόσβαση ούτε στις ε, χρηματαγορές ούτε στις ε, τραπεζικές αγορές διότι είναι πολύ μικρές επιχειρήσεις. Πρέπει λοιπόν να επικεντρώσουμε την δυνατότητα αυτή του θεσμικού πλαισίου ή ε, την ε, στήριξη ε, ενός συγκεκριμένου προβλήματος. Ήταν μεγάλη η πειρασμή που αντιμετωπίζαμε, αλλά πιστεύω ότι κάποια μέρα θα φτάσουμε σε μια ισορροπημένη κατάσταση και θα μπορέσουμε όχι μόνο με αριθμούς να παρουσιάσουμε τον πίνακα βαθμολόγηση των ε, κρατικών ενισχύσεων χωρίς να σας κάνουμε μία τελική αξιολόγηση διότι ακόμη δεν έχει έρθει ο χρόνος, είναι πρόωρο. Και ε, απαντώ τώρα στην ερώτηση της κυρίας ε, Γκουλάρ να προστατεύσουμε. Ε, στην αρχή έπρεπε να προστατεύσουμε, στην αρχή της κρίσεως, να προστατεύσουμε ό,τι ακόμη στεκόταν όρθιο. Τώρα όμως πρέπει να αλλάξουμε. Πρέπει να καταργήσουμε τις διαφορές ε, για να μπορούν να έχουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα έχουν ακόμη και του χρόνου πολλά προβλήματα. Πρέπει να τις βοηθήσουμε με ένα σύστημα το οποίο δεν θα είναι το ίδιο για όλους, υπό ορισμένες προϋποθέσεις αλλά δεν είναι πλέον χρόνος να πούμε ότι πρέπει να ε, προστατεύσουμε οτιδήποτε. Το 2011 σύμφωνα με το ότι διαβλέπουμε σήμερα από ότι θα είναι το 2011 από οικονομικής απόψεως χρηματοδοτήσεως πιστεύουμε ότι το 2011 θα είναι μια χρονιά όπου θα πρέπει να επιταχύνουμε τους ρυθμούς να υπάρξουν πολύ αυστηροί δημοσιονομικοί περιορισμοί να φύγουμε από την στρατηγική εκτάκτων κρίσεων χωρίς όμως να μπορέσουμε μπορέσουμε να πούμε ήδη ότι όλα έχουν επανέλθει στην τάξη και μας ξαναήρθε η παλιά καλή εποχή. Εκτός από την αναθεώρηση της άλλες πολιτικές οι οποίες καταρτίζονται ή θα καταρτιστούν, αυτό το οποίο συνέβη με τις γραμμές του Temporary Framework ήταν ότι οι συνθήκες της τακτικής εφαρμογής των προσανατολισμών κρατικών ενισχύσεων ε, ε, ε, επαρκούσαν. Δεν, δεν διέφεραν από το temporary framework. Οπότε ε, παρόλο που τα μέτρα αυτά αρχικά ήταν για το περιβάλλον ή για παρεμφερή, επειδή είμαστε εν πλήρη κρίση προσπαθήσαμε να χρησιμοποιήσουμε το καθεστώς φυσιολογικής κατάστασης και όχι έκτακτης κατάστασης. Νομίζω τέσσερις χώρες χρησιμοποίησαν αυτές τις γραμμές. Προς τον κύριο Πρεσέντο. Όταν όταν θα έρθει η ώρα θα αποσύρουμε ό,τι πρέπει να αποσυρθεί βάσει της ε, ε, πολιτικής αποφάσεως και πρέπει να σας πω ότι πριν το καλοκαίρι όταν συζητούσαμε με την Γενική Διεύθυνση και τις υπηρεσίες μας για να δούμε τι έπρεπε να γίνει με το προσωρινό πλαίσιο η πλειοψηφία ήταν ε, πιο αισιόδοξη όταν συζητούσαμε για να επανέλθουμε σε φυσιολογική κατάσταση κατάσταση το 2011. Αλλά μετά την κατάσταση της Ιρλανδίας είμαστε τώρα πιο προσεκτικοί και επιφυλακτικοί και από τις πληροφορίες τις οποίες λαμβάνουμε και εκτός Ευρωπαϊκής Ενώσεως δεν είμαστε τόσο αισιόδοξοι όσο είμαστε ε, με τη Γερμανία η οποία έχει αυτή την καταπληκτική εξέλιξη το δεύτερο εξάμεινο του 2010. Θα δούμε τι θα γίνει στην συνάντηση που θα έχουμε με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και να δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Μετά το καλοκαίρι έχει μειωθεί το, ε, Yo creo ε, ε, ε, αισιοδοξία μας σε σχέση, το, με, με το παρελθόν. Με συγχωρείτε που σας δίνω τόσους πολλούς αριθμούς, αλλά πολλά κράτη έχουν εφαρμόσει πολύ προσεκτικά προγράμματα. Χρησιμοποίησαμε 20% του ό,τι προσεφέρετο και θα μπορούσα να αναφέρω και δύο προβλήματα. Ελπίζω ότι θα έχουν ε, απαλληφθεί στις 31 Δεκεμβρίου με τις προσαρμογές τις οποίες θα κάνουμε. Ένα από τα προγράμματα, ε, προβλήματα αυτά ήταν ε, η ερμηνεία του προσωρινού πλαισίου συνδυάζοντας 500.000 ευρώ ανά επιχείρηση και τη δυνατότητα ενός επικουρικού δανείου. Υπήρχε μεγάλος κίνδυνος αλλά τώρα που θα διαγραφούν 500.000 στις 31 Δεκεμβρίου θα αλλάξουν τα πράγματα. Επίσης ε, υπήρχε μία χώρα και ίσως και δύο-τρεις ακόμη που κρυβόντουσαν έπρεπε να ε, διατυπώσουμε το προσωρινό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσαμε να στηρίξουμε τη βιομηχανία του κάθε κράτους. Τώρα έχουμε μόνο μία περίπτωση την οποία παρακολουθούμε για την κρατική ενίσχυση αλλά γενικώ πιστεύω ότι ο τρόπος εφαρμογής του προσωρινού προσωρινού πλαισίου ήταν σωστός και συμφωνώ με αυτά που είπατε για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις διότι ε, ε, όταν χρησιμοποιούνται ε, ενισχύσεις θα πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί αλλά να ξέρετε ότι το μήνυμά μου σαν επίτροπος για το 2011 είναι ότι θα πρέπει να προσαρμόσουμε αυτό το προσωρινό πλαίσιο και επιπλέον θα πρέπει να δούμε πώς χρησιμοποιούνται οι δημόσιοι πόροι τους οποίους χρησιμοποίησαμε κατά κόρον τα δύο τελευταία χρόνια. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τις ίδιες μεθόδους το 2011 και για να τελειώσει η κρίση δεν χρειάζεται μόνο μία φορολογική ολοκλήρωση, χρειάζεται και ανάπτυξη και για να υπάρξει ανάπτυξη πρέπει να ξεχάσουμε τις κρατικές ενισχύσεις, να αναθεωρήσουμε περισσότερο και να προσαρμόσουμε περισσότερο την ατζέντα του 2020. Ευχαριστώ. Τελειώνει ο χρόνος μας και έχω ακόμη τέσσερις ερωτήσεις, οπότε παρακαλώ να είστε όσο δυνατόν πιο σύντομοι. Ο Ντέρκ, ο και ο κύριος Σιμό. Ευχαριστώ. Οι κατευθυντήριε αρχέ για την αντιμετώπιση, γραμμέ για την αντιμετώπιση τη κρίση λέει ότι δεν πρέπει να υπάρχει αθέμητο ανταγωνισμό. Αν δείτε όμω την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών, οι, περιπτώσεις, ε, οι διάφορε περιπτώσει ε, διαφορετικά αντιμετωπίστηκαν. Για παράδειγμα, η ING κατηγορήθηκε για στρέβλωση του ανταγωνισμού με τη χρήση δημοσίου χρήματο, ενώ ε, κάμπεσέ και άλλε χώρε και άλλε τράπεζε όπω η Lloyds όχι. Δηλαδή, δόθηκαν ιδιαίτερες ε, εξουσίες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, περισσότερες από όσε είχε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, χρησιμοποιεί την πολιτική του ανταγωνισμού για να αναδιαρθρώσει και άλλους τομείς εκτός από τον οικονομικό ε, τομέα. Και το αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν ότι τελικά αντί να ε, παρεμποδίζει τον αθέμητο ανταγωνισμό, τον αυξάνει τελικά. Μήπως θα μπορούσατε λοιπόν να μας εξηγήσετε γιατί παρόμοιες περιπτώσεις αντιμετωπίστηκαν διαφορετικά και γιατί υπάρχει τόσο λίγη διαφάνεια. Θα ήθελα επίσης να πω μερισμένα πράγματα για τα προσωρινά μέτρα. Είπατε ότι θα εκπνεύσουν. Πόσο όμως είναι προσωρινό το προσωρινό αυτό πλαίσιο. Γιατί ο κύριος Τρισέ ήταν εδώ πριν από μία εβδομάδα και μας είπε ότι ε, και πάλι αρχίζουν να εισραίουν τα κεφάλαια ε, δεν, ε, και, ότι, αν οι κρατικές ενισχύσεις δεν καταργηθούν προοδευτικά θα αρχίσει η υπερβολική κεφαλαιοποίηση με αποτέλεσμα τελικά να έχουμε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Μια ερώτηση προς τους δύο επιτρόπους ομολογώ ότι εγώ έχω λίγο τρομάξει γιατί διαπιστώνω ότι υπάρχει μια Ευρώπη δύο ταχυτήτων. Βλέπω μπροστά μου ένα κομμάτι της Ευρώπης το οποίο ανακτά τις δυνάμεις της και με μεγάλη ταχύτητα. Και αυτό συμπεριλαμβάνει και το πιστοτικό ε, κομμάτι, το χρηματοπιστωτικό κομμάτι όπως το είπε και ο Γκαρσία Μαργκάλιο θα πρέπει να υπάρχει ζήτηση για πιστώσεις, αλλά η ζήτηση αυτή θα πρέπει να προέρχεται από αυτούς οι οποίοι μπορεί να επιστρέψουν τα χρήματα που θέλουν να δανειστούν. Οι μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχουν ξεκινήσει και προχωρούν ορισμένες χώρες ε, το κάνουν με διαφορετικές ταχύτητες. Θυμίζω ότι στην Ισπανία αυτά τα οποία γίνονται σε σχέση με τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας είναι ιδιαίτερα συγκεχημένα. Πιστεύετε ότι μήπως ότι αυτή η μεταρρύθμιση στην ουσία δεν είναι παρά ένα άλοθη, ο κύριος Κλίντς. Ευχαριστώ, αλλά η, ο κύριος Σαρκοζή είχε πει ότι θα πρέπει να βρεθεί παγκόσμια λύση στην παγκόσμια κρίση. Σήμερα όμως δύο χρόνια μετά από την αιχμή της κρίσεως πρέπει να σας πω ότι είμαι πολύ απογοητευμένος για τις αποφάσεις που ελήφθησαν διεθνώς, διότι είχαμε πει ότι όλες οι περιπτώσεις θα ρυθμίζονταν με τις ίδιες αρχές, τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης. Ο Πίτερ Σκίνερ τα έχει ε, εξετάσει και λέει ότι υπάρχουν περισσότερες διαφορές παρά κοινά σημεία. Επίσης ε, είπατε ότι θέλετε να βελτιώσετε την κατάσταση ε, των κεφαλαίων των τραπεζών χαιρόμαστε ε, που τίθεστε επικεφαλής αυτής της κινήσεως αλλά μετά οπισθοδρομείτε και ε, οι Ελβετοί βλέπετε ότι δεν συμφωνούν καν με τη Βασιλεία 2 και δεν θέλουν να εφαρμόσουν τη Βασιλεία 3 δηλαδή ε, κάθε απόφαση που λαμβάνετε μόνη της είναι, είναι λογική αλλά πρέπει να τα δούμε όλα αυτά μαζί και ε, να διαπιστώσουμε ότι ε, γίνεται πολύ πιο βαρύ το σύνολο και έτσι δεν μπορούμε να επιτύχουμε τον στόχο τον οποίο προσπαθούμε ε, να επιτύχουμε. Έχω μία ερώτηση, εδώ είμαι, σχετικά με την σημασία της προλήψεως και της προστασίας από την άλλη πλευρά, διότι είπατε ότι η πρόληψη είναι πάντοτε καλύτερη από τη θεραπεία. Αυτό όμως το οποίο θέλω να πω είναι ότι αν αναφερθούμε ε, στην νομοθεσία και το σημείο που αναφέρεται στο, στο θέμα αυτό βλέπουμε ότι υπάρχει προτίμηση για τα μέτρα θεραπείας δηλαδή να να απευθυνθεί κανείς στους καταθέτες όταν η τράπεζα καταρρεύσει αντί ε, να προλάβουν να καταρρεύσει η τράπεζα αυτή ε, και αυτό με το πρόσχημα του ανταγωνισμού με άλλες ε, τράπεζες οι ο οποίος θα πρέπει να υπερισχύσει. Όλα αυτά δεν βρίσκω να είναι συνεκτικά. Ο κύριος Αλμούνια. Δεν μπορείτε όμως να πάρετε το λόγο για τόσο πολλή ώρα όσο και προηγουμένως, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, μόνο πέντε λεπτά. Ακόμη λιγότερα θα χρειαστώ, κύριε Πρόεδρε. Για τον κύριο Επίνγκ. Για ποιο λόγο οι αποφάσεις για την ING, για την Credit Bank ή τη Lloyds ή οποιαδήποτε άλλη τράπεζα ε, δεν είναι ίδια. Γιατί είναι πολύ απλό. Δεν ήταν οι ίδιε περιπτώσει, ήταν διαφορετική η κατάσταση. Η εθνική αγορά για τον έναν, τον καλό ή τον κακό λόγο ε, είναι διαφορετικε Είναι διαφορετικε οι κατάστασεις, ε, οι χρηματοοικονομικέ ε, σε κάθε χώρα. Άλλο ε, ο, η χρηματοοικονομική αγορά στην Ολλανδία και άλλο αλλού. Είναι τελείω διαφορετικά στην Ολλανδία τα πράγματα από ό,τι στη Γερμανία, από ό,τι στη Γαλλία, από ό,τι στο Ηνωμένο Βασίλειο. Επομένω και οι αποφάσει είναι διαφορετικέ. Όμω είναι διαφανεί οι αποφάσει με την εξαίρεση των ε, στοιχείων εκείνων της απόφασης που για προφανείς λόγους δεν μπορούν να δημοσιοποιηθούν ε, γιατί θα στρεβλώσουν τελικά τον ανταγωνισμό Όμω υπάρχει μια ισότιμη μεταχείριση, όχι ταυτόσιμη, όχι ίδια, αλλά ισότιμη μεταχείριση και εμεί παρακολουθούμε την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών ε, με την ίδια αυστηρότητα και ε, πολύ στενά. Εγώ δεν είμαι υπεύθυνο για την βιομηχανική πολιτική. Ο Αντώνιο Τελιάνιο, ο συναδελφό μου, είναι υπεύθυνο για το θέμα αυτό. Απλώ δεν θα έπρεπε να υπάρχει κακή ερμηνεία για το τι θα πει σύγχρονη βιομηχανική πολιτική. Σύγχρονη βιομηχανική πολιτική, αποτελεσματική βιομηχανική πολιτική, δεν είναι τομεακή, ε, δεν... Ε, ε, δεν θέλουμε τίποτε άλλο εκτός από το να έχουμε οριζόντια μέσα για έναν ανταγωνιστικό βιομηχανικό τομέα και μια ανοιχτή οικονομία που μπορεί να ανταγωνιστεί ε, σε διεθνές επίπεδο. Τα μέσα ανταγωνισμού και στα αντιτράστ και στις κρατικές ενισχύσεις σκοπό έχουν αυτούς τους στόχους να εξυπηρετήσουν. Ενδεχομένως η έκθεση του Μάριο Μόντι για την εσωτερική αγορά να το αναφέρει καλύτερα. Ο ρόλος Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να υπάρχει μια ισχυρή εσωτερική αγορά για το 2020 και αυτό είναι που θέλουμε να επιτύχουμε. Αυτό χρειαζόμαστε άλλωστε. Προσωρινό θα πει προσωρινό. Σας το είπα και προηγουμένως. Το προσωρινό πλαίσιο όπως το γνωρίζαμε δεν θα εξακολουθεί να, από, να υφίσταται από 1η Ιανουαρίου του 2011. Κάποια στοιχεία όμως, κάποια στοιχεία θα εξακολουθούν να υφίστανται με τις προσαρμογές που θεωρούμε ότι χρειάζονται δεδομένων των συνθήκων, ε, ανάλογα με τις εταιρείες και φυσικά και σε σχέση με τις μικρομεσαίες ε, επιχειρήσεις. Οπότε, ναι, ξέρω πολύ καλά τι θα πει προσωρινό ε, και θέλω να πιστεύω ότι σε ένα μήνα ε, θα αλλάξουν ε, τα πράγματα για το 2011, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα, ώστε να προτείνουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να καταργήσει το προσωρινό πλαίσιο, αλλά δυστυχώς η επιθυμία αυτή, η ευχή αυτή μπορεί να μην πραγματοποιηθεί και μπορεί να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις και το επόμενο έτος και μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και πάλι κάποια εξαιρετικά μέτρα, όχι όμως τόσο εξαιρετικά και όχι τόσο εις όσο το 2009 και το 2010. Κύριε Τρεμόσα, η εποπτεία. θα είναι πολύ πιο αυστηρή χάρη στα μέτρα που ανέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Σεπτεμβρίου. Εάν το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο εγκρίνουν τα μέτρα αυτά, και ελπίζω αυτό να γίνει όσο το δυνατόν συντομότερα, τα μέσα αυτά θα είναι στη διάθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ Κανένα δεν τη τα είχε δώσει. Δηλαδή, ε, επαγρύπνηση, συντονισμό, ε, δημοσιονομικό και μακροοικονομικό συντονισμό. Πρόκειται για ένα πλαίσιο για την ε, στρατηγική από εδώ και στο εξή. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μας δίνουν τα μέσα αυτά και αυτή η επαγρύπνηση, να είστε βέβαιοι, θα είναι πολύ πιο αυστηρή από ό,τι ενδεχομένω εσείς να δεχόσασταν. Όμως πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε με τα μέσα αυτά πολύ καλή δουλειά. Κύριε ε, Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι βεβαίως πρέπει να περιορίσουμε το κίνδυνο και να αποφύγουμε να υπάρχει εποπτεία δύο ταχυτήτων και αυτό ισχύει για την εποπτεία τη δημοσιονομική αλλά και την ε, χρηματοοικονομική πρέπει να πω ότι η πρώτη ευθύνη για την δημοσιονομική εποπτεία βρίσκεται σε κάθε χώρα με τις σωστές αρχές. Αλλά εφ' θα υπάρχει και ένα πλαίσιο μιλήσαμε για το μεγάλο ραντάρ όπου οι εθνικές εποπτείες ε, θα ανταλλάσσουν τα πορίσματά τους ε, ε, με μία αλληλοεξάρτηση για να αποφύγουμε μία εποπτεία δύο ταχυτήτων και να μπορέσουμε να έχουμε μία ενιαία αγορά και όχι δύο ταχυτήτων και αυτός είναι ο στόχος της ε, ανάπτυξης την οποία ε, προσβλέπουμε για την ε, εσωτερική αγορά για να μπορέσει να υποφεληθεί ο καθένας και ο καταναλωτής και γι' αυτό προσπαθώ και εγώ να προωθήσω την πολιτική συνοχής την οποία επενόησε η δίκηση Ντελόρ για να αποφύγει εδαφικές, εδαφικούς περιορισμούς ε, σε ένα σύνολο της κοινότητος. Ε, γι' αυτό και πρέπει να λάβουμε τα σωστά μέτρα τώρα παρακολουθώντας τι γίνεται από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού δεν πρέπει να ξεχνάμε την Κίνα, την Ινδία και άλλες περιοχές των οποίων οι αρχηγοί κρατών έχουν προσυπογράψει τα μέτρα του G20 και ακόμη και αν αυτή τη στιγμή υπάρχει ακόμη μια εντεπαράθεση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης αυτό στο μέλλον θα μειώνεται συνέχεια Υπάρχουν περισσότεροι στο G20. Εγώ όμως δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος όσο εσείς. Δεν πρέπει να είμαστε αφελείς, αλλά δεν πρέπει να προσάπτουμε λανθασμένες προθέσεις τους Αμερικανούς, διότι οι Αμερικανοί εφαρμόζουν τα μέτρα που αποφασίσαμε όλοι μαζί στο G20. Έχουν ψηφίσει μία νομοθεσία χιλιάδων 4.000 σελίδων που θα χρειαστεί χρόνια να εφαρμοστεί. Εμείς έχουμε ε, στιγμιές οδηγίες και κανονισμού αλλά μέσα σε ένα πλαίσιο που σας παρουσίασα πέρυσι τον Ιούνιο. Επίσης το τραπεζικό μας σύστημα δεν μοιάζει με το αμερικανικό και είμαστε σε στενή σύνδεση συχνά διότι έχω συνεργαστεί με τους Αμερικανούς επόπτες για τα χρηματοοικονομικά παράγωγα για να καταλήξουμε ε, στις ίδιες μεθόδους. Με τον κύριο Γκάιτνερ και τους συνεργάτες τους συμφωνήσαμε ότι θα εφαρμόσουν την ε, βασιλεία 2 προς 3 στα μέσα του επομένου έτου ε, για να ε, υπάρχει ένας παραλληλισμός μεταξύ μας. Βέβαια πρέπει να προσέξουμε κάτι πάρα πολύ. Καταρχήν ε, την, την τρίτη, το, την Βασιλεία Τρία και την εφαρμογή της, δηλαδή τους αναλογιστικούς ε, κινδύνους, ε, διότι πρέπει οι Αμερικανοί να συμμορφωθούν στις δεσμεύσεις που ανέλαβαν μαζί μας σχετικά με ε, τη Βασιλεία. Και επίσης κάτι που πρέπει να συμφωνήσουμε είναι οι λογιστικοί κανόνες. Ε, όταν λοιπόν βλέπει κανείς από πού ξεκίνησε κύριε Κλίνς βλέπετε ότι υπάρχει μία πρόοδος, υπάρχει μία παγκόσμια διακυβέρνηση με κάποια αξία ε, και βασίζεται σε αποφάσεις που έχουν ληφθεί από κοινού. Δεν υπάρχει ένα μόνο μέτρο το οποίο θα μπορέσει να προστατεύσει τους καταθέτες και ε, τους αποταμιευτές αλλά ε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μία εγγύηση για τους καταθέτες και τους αποταμιευτές και επίσης ε, θα πρέπει ε, να έχουμε ένα σύστημα συνεκτικό που να ισχύσει και στην Αυστρία ακόμη διότι εκεί υπήρχε μία, ένα διαφορετικό σύστημα αλληλασφαλίσεως των κινδύνων όπου οι μεν βοηθούσαν τους άλλους αλλά ε, υπάρχουν εχέγγυα και προς τους καταθέτες και τους αποταμιευτές και όλα αυτά πρέπει να συνδυαστούν με την εξωτερική εποπτεία, την εσωτερική εποπτεία, την καλή διακυβέρνηση, τα μέτρα επεμβάσεως, ένα σύνολο δηλαδή που μπορεί να βοηθήσει ή να προστατεύσει επαρκώς τους καταθέτες και τους αποταμιευτές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και για τα μέλη και τα μέλη για τις εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ερωτήσεις. Θα περάσουμε στο δεύτερο τμήμα. Θα υπάρξει ένα διάλειγμα τριών-τεσσάρων λεπτών μόνο για να έρθουν εδώ οι νέοι ομιλητές και να εγκατασταθούν. Okay, Καλώς. Θα συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Περνάμε στις απόψεις τώρα πλέον των ε, συμμετεχόντων στις αγορές. Τέσσερις θα είναι οι ομιλητές. εκπρόσωπος Σάιντσαβάντ της Σανταντέρ, ε, της ε, εταιρείας Σανταντέρ. Ε, Παρακαλώ πέντε λεπτά και μην ξεπεράσετε το χρόνο σας κύριε Πέρες Ρενοβάλες. Θα ήθελα καταρχάς ε, να σας εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου που μας δίνετε τη δυνατότητα να παριστάμεθα εδώ σήμερα εκ μέρους του ομίλου Σανταντέρ και να μιλήσουμε για ένα από τα ζητήματα που βρίσκονται υπό συζήτηση αυτή τη στιγμή. Παρακολουθούμε όλες τις ε, μεταρρυθμίσεις που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ε, είμαστε πολύ ευγνώμονες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί στην Επιτροπή σας που μας κάλεσε να είμαστε εδώ σήμερα. Λέγομαι Πέρες Ρενόβαλες, ε, είμαι αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και Νομικός Διευθυντής της Banco Santander και θα ήθελα πριν μπω στο θέμα να σας παρουσιάσω την τράπεζα που εκπροσωπώ. Είναι ένας όμιλος ε, λιανικής εμπορικής τραπεζικής. Έχουμε σημαντική παρουσία σε εννέα κύριες αγορές ε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία, Γερμανία και ε, Ηνωμένε Πολιτείε και Λατινική Αμερική με ιδιαίτερη παρουσία στη Βραζιλία. Ήμασταν ε, πολύ ανθεκτικοί κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης, που σημαίνει ότι είναι μία, ένα από τα μεγάλα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δεν χρειάστηκε άμεση κρατική ενίσχυση. Και αυτό φάνηκε και από τα αποτελέσματα των προσφάτων ε, τεστ αντοχών που έγιναν από τους Ευρωπαίους επόπτες. Και τα ισχυρά μας θεμέλια ε, και από απόψε ως ε, ε, αλλά και ισολογισμού μας επέτρεψαν και αυτόνομα αλλά και με εξαγορές να αναπτυχθούμε. Παράδειγμα αυτής της ανάπτυξης είναι η εξαγορά της Alliance and Leicester και τμήματων των Bradford and Bingley και της Royal Bank of Scotland στο Ηνωμένο Βασίλειο η Λιανική Τράπεζα της SEB στην Γερμανία και προσφάτως ε, η εξαγορά του 70% περίπου της Bank Sachodny VBK στην Πολωνία. Όλο το μετοχικό κεφάλαιο θα εξαγοράσουμε τελικά, γιατί θα υπάρξει ένας διαγωνισμός ε, και εμείς θα προτείνουμε να λάβουμε το 100%. Εκτός λοιπόν ε, από τα ε, περιουσιακά αυτά στοιχεία τα οποία θα εξαγοράσουμε, Εξαγοράσαμε τράπεζες οι οποίες διαφορετικά ε, θα είχαν χρειαστεί κρατική ενίσχυση και έτσι εμείς ενισχύουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και ενισχύουμε και την οικονομική σταθερότητα. Θα ήθελα να περάσω τώρα στο θέμα της σημερινή ακρόασης. Τρία σημεία θα ήθελα να φέρω σε σχέση με το, τους προσωρινούς κανόνες κρατικής ενίσχυσης. Ε, που εγκρίθηκαν για την κρίση. Πρώτον, ήταν μια εξαιρετική κατάσταση ε, η κρίση που όπως είπε και ο Επίτροπος Αλμούνια χρειάστηκε εξαιρετικά μέτρα για την ενίσχυση της σταθερότητας του χρηματοοικονομικού συστήματος και την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαδραμάτισε το ρόλο της ε, γιατί έθεσε προσωρινές διαδικασίες και αντιμετώπισε πολλές περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων. Για παράδειγμα, σχέδια αναδιάρθρωσης και περιορισμούς δραστηριοτήτων των ιδρυμάτων που είχαν λάβει κρατική ενίσχυση. Και επίσης έκαναν και σημαντικές ε, έρευνες ε, οι υπηρεσίες Ευρωπαϊκής Επιτροπής όποτε αυτό χρειαζόταν. Κατά τη διάρκεια της κρίσης διαπιστώσαμε ότι η αποζημίωση του ισρεόμενου ε, του κεφαλαίου ήταν κάτω από τις τιμές αγοράς. Ε, όταν δεν υπήρχε χρονικός περιορισμός για την αποζημίωση ή δεν υπήρχαν όροι ε, για τη διαφάνεια, είδαμε ότι σε μερικές μόνος περιπτώσεις η διανομή των μερισμάτων στου μετόχου μετόχους έλαβε χώρα. Γι' αυτό πιστεύουμε ότι η κρατική ενίσχυση πρέπει να δίδεται από του εξή όρου. Πρώτον, πρέπει να περιορίζεται σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ε, είναι βιώσιμα. Επίση, ε, η αξιολόγηση των μέσων ε, πρέπει να γίνεται επί τη βάση των τιμών τη αγορά. Πρέπει να είναι προσωρινή και να περιλαμβάνει κίνητρα για να αποζημιώσει το ίδρυμα το κράτο. Και επίση πρέπει να είναι διαφανή και να υπόκειται σε όρου. Το δεύτερο σημείο που θα ήθελα να είναι ότι παρά το γεγονό ότι είναι σημαντική η κρατική ενίσχυση για την οικονομική σταθερότητα, πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά τι στρατηγικέ εξόδου και να καταρτήσουμε σχέδια για την επιστροφή στις, ε, σε κανονικότητα. Δηλαδή, να περάσουμε σε καιρό ειρήνη, ε, για να το πούμε έτσι. Αυτό σημαίνει και ε, εξόφληση της κρατικής ενίσχυσης, αλλά και ε, ιδιωτικοποίηση και πάλι ορισμένων ε, ιδρυμάτων. Όσο διατηρείται η κρατική ενίσχυση, τόσο υπάρχει μεγαλύτερο κίνδυνο κίνδυνος στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Γιατί πολλές φορές είναι χαμηλότερο το κόστος ε, της ε, κυβερνητικής εγγύησης και δεν είναι ισότιμο το πεδίο συναλλαγών. Ε, αυτό το ζητούμε από το Δεκέμβριο του 2008, εξακολουθούμε να το ζητούμε και σήμερα και γι' αυτό χαιρετίζουμε τα νέα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εγκρίθηκαν τον Ιούλιο του 2010 και τα οποία ενέκρινε και το Συμβούλιο Κοφήν. Το τελευταίο και, το τρίτο και τελευταίο σημείο που θα ήθελα να θίξω έχει να κάνει με το μέλλον. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν ε, τα θεμέλια του χρηματοπιστωτικού συστήματος και να μειώσουμε την πιθανότητα επανάληψης της οικονομικής κρίσης. Οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να διασφαλίσουν ότι σε μελλοντική κρίση αν υπάρξει και δεν μπορούμε να την αποφύγουμε για οποιοδήποτε λόγο, ότι δεν, υπάρχει λόγος, δεν θα υπάρχει λόγο προσφυγής στην κρατική ενίσχυση. Πέντε βασικοί τομείς μεταρρύθμισης ε, πρέπει να ε, γίνουν για την ενίσχυση του οικονομικού συστήματος. Πρώτον, το κεφάλαιο χρειαζόμαστε καλύτερο λόγο κεφαλαίου, καλύτερη ποιότητα λόγο κεφαλαίου, δηλαδή οι απαιτήσει κεφαλαίου πρέπει να συνδέονται με κίνδυνο, επομένω, όσο μεγαλύτερη είναι η άλψη κινδύνου, τόσο περισσότερο κεφάλαιο να ε, έχουν τα ιδρύματα αυτά. Το θέμα της ρευστότητας. Πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ρευστότητα ώστε να επαφιέμεθα, να εξαρτώμαστε λιγότερο από χονδρική χρηματοδότηση. Επίσης, εταιρική διακυβέρνηση. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να έχουν ε, ανεξάρτητη ε, διαχείριση κινδύνου και τα διοικητικά συμβούλια πρέπει να παρακολουθούν ε, το σχεδιασμό και την εφαρμογή των ε, πολιτικών αποζημίωση. Διακόπτη πρόεδρο. έχετε ακόμη δύο λεπτά. Καλύτερα να ολοκληρώσετε γιατί έχετε, έχετε ξεπεράσει το χρόνο σας. Um, Ζήτησα συγγνώμη από τον ομιλητή, αλλά έπρεπε να διακόψει γιατί αλλιώς δεν θα υπήρχε χρόνο ερωτήσεων. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Βίνκ από την ING. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Εμείς ε, προσκληθήκαμε να συμμετέχουμε στη σημερινή συνεδρίαση και νομίζω ότι είναι σημαντική πρωτοβουλία της Επιτροπής Οικονομικών ε, και Νομισματικών Θεμάτων και με χαρά η ING θα συμμετέχει. Ε, λάβαμε κρατική ενίσχυση για να αντιμετωπίσουμε τις συνέπειες ε, των προβλημάτων που αντιμετωπίσαμε στο θέμα των χαρτοφυλακίων των, υποθηκών σε, ένα, σε μια αγορά χωρίς ρευστότητα και ζητήθηκε από την ING να μειώσει τον ισολογισμό τη κατά 45%. Επίσης ε, τέθησαν κάποιοι όροι από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή που περιορίζουν τη συμπεριφορά μας για τρία χρόνια. Όπως γνωρίζετε, εμείς έχουμε καταθέσει προσφυγή στο Γενικό Δικαστήριο του Λουξεμβούργου για κάποια στοιχεία της ε, απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και επειδή εκρεμεί η υπόθεση δεν μπορώ να μπω σε πολλέ λεπτομέρειες για ε, μερικά ζητήματα. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η χρηματοπιστωτική κρίση ήταν άνευ προηγουμένου κατάσταση που επιζήτα ακόμη και τώρα ε, εξαιρετικές παρεμβάσεις. Ε, πραγματικά πρέπει να αναγνωρίσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την άμεση ανταπόκρισή της. Ε, το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων για τον χρηματοπιστωτικό τομέα έδωσε στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να δώσουν ενίσχυση στις τράπεζες για τη διατήρηση του χρηματοπιστωτικού τομέα, ενώ παράλληλα προστάτευσε την εσωτερική αγορά. Δυστυχώς, τη στιγμή της κρίσης δεν ε, υπήρχε πανευρωπαϊκή δυνατότητα κρατικής ενίσχυσης. Κάθε κράτος μέλος έπρεπε να αντιμετωπίσει τις συνέπειες ε, με, το δικό της τρόπο και αυτό σημαίνει διαφορετικές προσεγγίσεις ε, στα διάφορα κράτη-μέλη. Σήμερα λοιπόν θα ήθελα να δείξω τρία ζητήματα που ενδεχομένως να θέλει να εξετάσει μεγαλύτερη λεπτομέρεια το Κοινοβούλιο και συγκεκριμένα η αρμόδια επιτροπή σας. Πρώτον, υπήρξαν κάποιες, ε, κάποιοι περιορισμοί ε, στη συμπεριφορά της τράπεζάς μας ε, και πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτό επιτρέπει να εξακολουθεί να υφίσταται ένα ισότιμο πεδίο. Κάτι που πρέπει να αναλύσουμε περισσότερο είναι κατά πόσο οι δεσμεύσει αυτέ, οι περιορισμοί ε, συμπεριφορά και αναδιάρθρωση ε, είναι επικερδεί για την εσωτερική αγορά, ε, για τον ανταγωνισμό και του καταναλωτέ. Γιατί μερικέ φορέ μπορεί να έχουμε αθέμητο ανταγωνισμό, όπω για παράδειγμα το price leadership, δηλαδή απαγόρευση χρήση του δημοσίου χρήματο με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. Αυτό μπορεί τελικά να μην εξυπηρετεί τι ανάγκε πραγματική οικονομία και των καταναλωτών. Επίση, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι ο στόχο του ισότιμου ε, πεδίου, τη ισότητα, ε, ε, επιτυγχάνεται με τη σωστή βαθμονόμηση όταν ε, γίνεται σύγκριση των διαφορετικών πτώσεων κρατικής ενίσχυσης. Για παράδειγμα, στήριξη ρευστότητα των τραπεζών είναι κάτι που δεν συμπεριλαμβάνεται στην αξιολόγηση συγκρισιμότητα τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, ενώ τα μέτρα ανακεφαλαιοποίηση και εγγυήσεων συμπεριλαμβάνονται. Επίση, τα εθνικά προγράμματα στήριξη ε, σε ορισμένε χώρε ε, δεν συνάδουν με το πνεύμα της εσωτερικής αγοράς ο μόνος τρόπος να υπάρχει ισότητα είναι η άμεση και έμεση κυβερνητική στήριξη να συμπεριλαμβάνεται στην αξιολόγηση. Επίσης, μεγάλη σημασία και στο πλαίσιο της κρατικής ενίσχυσης είναι και το IFRS, ε, τα λογιστικά πρότυπα δηλαδή και η οδηγία για, τα, για τις ε, απαιτήσει κεφαλαίου να ε, εφαρμόζονται με συνέπεια σε όλη την Ευρώπη, αλλιώς καταλήγουμε σε στρέβλωση του ανταγωνισμού. Είναι επίση σημαντικό ε, να, ο στόχο τη ισότητα να μην αξιολογείται μόνο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά να λαμβάνει υπόψη το παγκόσμιο πλαίσιο στο οποίο ανταγωνίζονται οι τράπεζε. Η ευρωπαϊκή οικονομία χρειάζεται ανταγωνιστικούς παίκτε ε, στην παγκόσμια αγορά για να ανταγωνίζεται με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε χώρε όπω οι ΗΠΑ και η Κίνα. Πιο συγκεκριμένα, απαιτήσει αναδιάρθρωση και ε, περιορισμοί μεγάλη εμβέλεια επιβλήθηκαν στι τράπεζε Ευρωπαϊκή Ένωση, εντό Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και ε, έλαβαν σημαντικά ε, σημαντική κρατική ενίσχυση ε, και άλλες, ε, και άλλες τράπεζες που δεν έλαβαν δεν έχουν να αντιμετωπίσουν αυτό το βάρος. Μια πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι εντελώς μεμονωμένη σε ένα πεδίο ανταγωνισμού παγκόσμιο δεν εξυπηρετεί τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε της πραγματικής οικονομίας. Κάτι που με οδηγεί στο δεύτερο, μου, ε, στο δεύτερο θέμα που θα ήθελα να θέσω, την ε, ανάγκη αξιολόγηση κρατικής ενίσχυσης ε, για να αξιολογήσουμε πόσο είναι διαφανή και προβλέψιμα τα αποτελέσματα. Έχει διοικητική ευχέρεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την εφαρμογή των κατευθυντηρίων γραμμών, ε, όμως αυτό αναθεωρείται εκ των υστέρων από τα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Πρέπει να υπάρξουν κατευθυντήριες γραμμές, περισσότερο λεπτομερείς, προκειμένου να διασφαλιστεί ε, συνεπέ συγκρίσιμο, συνεπές και προβλέψιμο αποτέλεσμα της αξιολόγηση Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πιστεύουμε λοιπόν ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το θέμα των κρατικών ενισχύσεων τα τελευταία δύο χρόνια πρέπει να αναλυθεί περισσότερο, να αναθεωρηθεί και όταν χρειάζεται να βελτιωθεί. Μελλοντική βελτίωση του πλαισίου πρέπει να εφαρμόζεται για όλε τι τράπεζε που έλαβαν κρατική ενίσχυση για να υπάρχει ένα πεδίο ισότητα στο πλαίσιο τη εσωτερική αγορά. Και έτσι φτάνω στο τρίτο σημείο που θα ήθελα να θίξω και είναι και η τελευταία μου παρατήρηση που είναι το ζήτημα κατά πόσο θα έπρεπε να παραταθεί το προσωρινό πλαίσιο. Δεδομένου ότι η ανάκαμψη μόλις άρχισε και είναι ακόμη ευαίσθητη, επίσης διαφέρει από χώρα σε χώρα, πιστεύουμε ότι είναι προς συμφέρον όλων να παραταθεί το προσωρινό πλαίσιο για κάποιο χρονικό διάστημα. Τα διδάγματα από τα τελευταία δύο χρόνια μπορούν να μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε το πλαίσιο αυτό. Επίσης, υποστηρίζουμε πλήρως ε, τις ε, τρέχουσες νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα μειώσουν την ανάληψη κινδύνου και θα ενισχύσουν την συνολική σταθερότητα του χρηματοοικονομικού συστήματος. Κυρία Πρόεδρε, θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντας ότι θεωρούμε σημαντικό να υπάρξουν διαβουλεύσεις για την αναθεώρηση του προσωρινού πλαισίου, γιατί αυτό θα επιτρέψει στα στα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λάβουν υπόψη τις απόψεις όλων των εμπλεκομένων φορέων. Σας ευχαριστώ πολύ. Φανώ σε πέντε λεπτά είναι δύσκολο να σταματήσει κανείς. Θα ακούσουμε τώρα τον υπεύθυνο αναλυτή της ε, Κεντρικής Τράπεζας της Ιταλίας. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε το λόγο. Θα ήθελα να διευκρινίσω ορισμένα πράγματα. Τα τελευταία δύο χρόνια είχα πάρει μέρος σε ένα πρόγραμμα κοινό ανάμεσα στην ε, Banca d'Italia και την ε, Τράπεζα Διεθνών Διαφετήσεων για να βρούμε μέτρα υποστήριξης του ε, πιστοτικού τραπεζικού συστήματος έχω συγκεντρώσει την προσοχή μου σε θέματα ε, εγγυήσεων ε, ε, ομολόγων τραπεζικών, κρατικών εγγυήσεων, αλλά παρόλα αυτά οι απόψεις τις οποίες θα εκφράσω είναι θα έλεγα προσωπικές. Η παρουσίασή μου λοιπόν θα καλύψει δι, τρεις θα έλεγα περιπτώσεις Καταρχάς θα μιλήσω για το μέγεθος και την αποτελεσματικότητα των κρατικών εγγυήσεων στον τομέα της έκδοσης τραπεζικών ομολόγων, να μιλήσω για τις τρευλώσεις που πιθανώς μπορεί να δημιουργήσει μια τέτοια παρέμβαση και τρίτο να δούμε πού βρισκόμαστε σήμερα, αν οι εγγυήσει αυτές δηλαδή θα πρέπει να επεκταθούν και για το 2011. Να μιλήσω λίγο για το μέγεθος και την αποτελεσματικότητα αυτών των μέτρων σε εισαγωγικά διάδοσης, διάσωσης, του χρηματοπιστωτικού τομέα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος της Banca d'Italia και της Διεθνούς Τράπεζας Διευθετήσεων έγινε η ανακοίνωση των μέτρων κατά τη διάρκεια του 2008. Οι ανακοινώσεις αυτές πράγματι βοήθησαν για να αποφύγουμε θα έλεγα το σενάριο της χείριστης μορφής, της χείριστης περίπτωσης, αυτό το είπε και ο Επίτροπος Σαλμούνια και συμφωνούμε μαζί του, τα μέτρα αυτά στην ουσία βοήθησαν να υπάρξει τροφοδοσία σε, ε, σε χρηματοδοτήσεις για τις ε, τράπεζες, ιδιαίτερα στον τομέα ε, των ομολόγων. Νομίζω λοιπόν ότι η παρέμβαση εκεί υπήρξε αποτελεσματική σχετικά με τις εγγυήσεις για τα ομόλογα τα τελευταία 2-2,5 χρόνια. Να πω ότι μέχρι τα μέσα του 2009 το ποσοστό εκδόσεων ήταν πάρα πολύ υψηλό, μετά υπήρξε μια μείωση των εκδόσεων ομολόγων και των εγγυήσεων που δόθηκαν προς την κατεύθυνση αυτή. Υπήρξαν δύο κορυφώσεις βέβαια φέτος τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο και αφορούν ουσιαστικά ένα μεγάλο πιστοτικό ίδρυμα σε μία χώρα κάθε φορά. Τώρα για το δεύτερο σημείο είναι οι στρεβλώσεις που μπορεί να προκαλούν οι εγγυήσει αυτές. Οι εγγυήσει αυτές, τα τραπεζικά ομόλογα, αυτό το οποίο είδαμε τελικά είναι ότι στην ουσία οδήγησαν στο κόστος δανεισμού των τραπεζών να μην αντικατοπτρίζει, θα έλεγα, την πιστοτική αξία των τραπεζών αυτών και την πιστοληπτική τους ικανότητα, αλλά την πιστοληπτική ικανότητα του κράτους που εκδίδει τις εγγύησεις. Αυτό έχει κάποιες ε, περιπλοκές κάποιες αδύναμες τράπεζες οι οποίες έχουν όμως ένα ισχυρό εγγυητή δανείστηκαν θα έλεγα πολύ ακριβά ενώ κάποιες ε, υγιείς οικονομικά τράπεζες ε, που δεν είχαν πίσω τους μια ισχυρή χώρα δανείστηκαν πιο ακριβά. Μια δεύτερη ομάδα στρεβλώσεων θα έλεγα είναι ότι οι μεγάλες τράπεζες πήραν τη μερίδα του λέοντος πρώτες. Αυτή ήταν η κατάσταση σε διάφορες ε, χώρες. Και αυτό το οποίο επίσης παρατηρήσαμε είναι ότι ήδη από το 2009 που σταθεροποιήθηκαν οι αγορές κάπως και οι εντάσεις κατέβηκαν, η πιστοληπτική ικανότητα των χρηστών των εγγύσεων αυτό έχει χαμηλώσει. Δηλαδή ε, η αξιολόγηση, η πιστοληπτική των τραπεζών κατέβηκε από τον μέσο όρο ε, που είχαμε πριν από το 2009. Αυτό σημαίνει ότι οι εγγυήσει αυτές στην ουσία οδήγησαν στην αναβολή κάποιων μεταρρυθμίσεων που ήταν απαραίτητες για ένα χρονικό διάστημα. Έχουμε λοιπόν κάποιες τρευλώσεις από τις κρατικές εγγυήσει. Επηρέασαν και τον ανταγωνισμό. Υπήρξε στρέβλωση ουσιαστικά του ανταγωνισμού. Υπήρξε μια κακή μάλλον χρήση των διαθεσίμων πόρων και αυτό θα επηρεάσει μακροπρόθεσμα την παραγωγικότητα του πιστοτικού τομέα. Θα ήθελα να αναφερθώ στο τρίτο και τελευταίο τμήμα. Α, θα πρέπει να διευρύνουμε τις εγγυήσει χρονικά στο 2011. Η απάντηση είναι βασικά ναι. Αν και η χρήση των εγγυήσεων αυτών και η ζήτηση έχει μειωθεί από τα μέσα του 2009, νομίζω ότι η διεύρυνση για το 2011 είναι χρήσιμη για δύο λόγους βασικά. Πρώτον, ότι η αναχρηματοδότηση ομολόγων από τις τράπεζες έχει ήδη ξεκινήσει. Αυτές οι ε, ανάγκες αναχρηματοδότησης στην ουσία χαρακτηρίζονται από υψηλό διαφορετικό κίνδυνο και από την άλλη στα πλαίσια της αγοράς η οποία αυτή τη στιγμή εξακολουθεί να είναι ε, όχι ιδιαίτερα εύρυθμη. Τον προηγούμενο Ιούλιο η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε κάποια θα έλεγα πιο αυστηρά κριτήρια σε σχέση με τη χορήγηση των εγγυήσεων και αυτές οι εγγυήσει σίγουρα λειτουργούν μειωτικά για τις τρευλώσεις τις οποίες προαναφέρθηκα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Τώρα προχωράμε στον κύριο Ρόλντ Κάρτον ε, ο οποίος ε, ε, είναι μέλος ε, της ομάδας αντιτράς και συνδεγονισμού. Ευχαριστώ που με καλέσατε σήμερα εδώ να βοηθήσω και να συμμετάσχω στην Επιτροπή σας και θα αναφερθώ εις ε, την εταιρεία μου που καλύπτει την Ευρώπη, ε, την Μέση Ανατολή και τον Περσικό κόλπο ε, και την Ασία και έχουμε συμμετάσχει εις τα μέτρα αναδιάρθρωσης για λογαριασμό πελατών μας. Θα σας πω λοιπόν τι γίνεται σήμερα χρησιμοποιώντας το Wii όπως το χρησιμοποιούσε η Βασίλισσα Βικτόρια ε, και αυτό που θα σας παρουσιάσω δεν ε, θα είναι η άποψη της Βασίλισσας Βικτορίας αλλά ε, ούτε προσπαθούμε να προωθήσουμε τα εμπορικά συμφέροντα οποιοδήποτε μέλους της εταιρείας. Είχαμε αναλάβει τεράστιες προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανταποκρίθηκε και σαν θεσμικό όργανο και σαν ομάδα πολύ προσιλωμένων ατόμων. Προσπαθούμε ε, να ε, αναδιαρθρώσουμε, ε, να συμβάλλουμε στην αναδιάρθρωση την οποία επιζητά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία ζητά ευελιξία και διακριτικότητα στη λήψη αποφάσεων σε μεμονωμένες περιπτώσεις κατά τρόπον ώστε να υπάρξει μία συνεκτική πολιτική για όλο το προσωρινό πλαίσιο και ε, βλέπουμε ότι η ευρωπαϊκή πολιτική έχει χρησιμοποιήσει ευελιξία για την ε, επίλυση των διαφόρων περιπτώσεων διότι όπως είπε ο κύριος Σαλμούνια κάθε τράπεζα και κάθε περίπτωση διαφέρει. Προσπαθούμε λοιπόν ε, να διατυπώσουμε τις συνθήκες ε, μη ενός προγράμματος αναδιάρθρωσης και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην περίπτωση προσπαθεί ε, να ε, εφαρμόσει μία απόφαση η οποία συνάδει με τις προηγούμενες αποφάσεις της παρόλο που κάθε κράτος έχει τις ιδιομορφίες του και κάθε τράπεζα έχει τις δικές της. Ε, όσον αφορά την ευελιξία και ε, την διάκριση ε, υπάρχει η αντιμετώπιση των προθεσμιών που καθορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροφή για τις επανιδιωτικοποιήσεις, τις πωλήσει και άλλων διαρθρωτικών μέτρων τα οποία θα εφαρμοστούν στην αγορά για τα επόμενα έτη και βλέπουμε ότι ενδέχεται να μην υπάρχουν πολλοί οι δυνητικοί αγοραστές με μεγάλες δυνατότητες. Οι τιμές λοιπόν είναι χαμηλές και η υποπίεση πωλήσει μπορεί να εμποδίσουν την επιβίωση της τράπεζας και για σας ε, ε, επίσης πρέπει κανείς να λάβει κανείς υπόψη του την ε, βιωσιμότητα και τον κίνδυνο για τον φορολογούμενο. Οπότε το κράτος μέλος θα πρέπει εφόσον το, το κράτος επιδεικνύει καλή διαγωγή ε, να οδηγήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξασκήσει μεγαλύτερη ευελιξία για να μπορέσει να κλείσει την πόλη ε, την πόρτα του άρθρου 107.3β. Το τρίτο σημείο μας αναφέρεται στην ε, διαφάνεια της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι η διαφάνεια χρειάζεται και ιδιαιτέρως χρήσιμη για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης ε, ιδίως όταν πρόκειται ε, για μεμονωμένες περιπτώσεις. Ξέρουμε ότι αυτό το έργο είναι πολύ δύσκολο ιδίως διότι το πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων απαιτεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προσεγγίσει ε, την ανάλυση της με πολύ αυστηρά μέτρα αλλά χρειάζεται συγχρόνως και επιστημονικές γνώσεις για να μπορέσουμε να μεγιστοποιήσουμε την διαφάνεια σε κάθε δεδομένη περίπτωση και έτσι κατά λίγο στο τελευταίο επιχείρημά μου όπου συμφωνούμε με την κυρία Γκουλάρ, τον κύριο Γκαρσία και την κυρία Ίντφελτ που είπαν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Κομισιόν θα πρέπει να κάνουν έναν απολογισμό των μέτρων που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι τώρα για να βεβαιωθούμε ότι ήταν επιτυχή, δηλαδή συνδύασαν τους ηθικούς κινδύνους, την στήριξη των τραπεζών, την αποφυγή στρεβλώσεων και την αποφυγή των δυσμενών επιπτώσεων, έστω και άθελα στην πραγματική οικονομία και με αυτό το σχόλιο τελειώνω. Ευχαριστώ. Θα συνεχίσουμε τις συζητήσεις τώρα και τις ερωτοαπαντήσεις. Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ζήτησαν το λόγο, αλλά οι επίτροποι ε, μίλησαν για αρκετή ώρα και δεν θα τους δώσω το λόγο, εκτός και αν στο τέλος έχουμε κάποιο επιπλέον χρόνο. Στον κατάλογό μου έχω αρκετούς συναδέλφους Λοιπόν, ε, κάθε ερώτηση θα την χάνει απαντήσεων. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να θέσω μία ερώτηση προς τον κύριο Κάβλτον και τον κύριο Λεβί. Τώρα πολύ σωστά είπατε για την ανάγκη που υπάρχει να επιδείξουμε μία κάποια ευελιξία αλλά και υψηλή διακριτικότητα στα πλαίσια της αξιολόγησης των εμπλεκομένων στην προσπάθεια επίλυσης της κρίσης. Από την άλλη, αυτό θα μπορούσε ε, να οδηγήσει σε κάποιες ε, άδικες αντιμετωπίσεις ορισμένων από τους ε, εμπλεκομένους και να στρεβλώσει τον ανταγωνισμό και θα ήθελα τα σχόλιά σας για το τι θα λάβετε υπόψη έτσι ώστε να διασφαλίσετε την ίση μεταχείριση των εμπλεκομένων από τις αρχές. Ακούγοντας αυτά τα οποία είπε ο κύριος Πέρες Ρενοβάλες, είδα ότι μπορούμε να μιλήσουμε για μια δίκαιη αντιμετώπιση των εμπλεκομένων μόνο στα πλαίσια των κρατικών βοηθειών, ενισχύσεων. Μήπως όμως κάτι τέτοιο θα πρέπει να λάβει υπόψη και τα προγράμματα αναδιάρθρωσης, όχι μόνο ευρωπαϊκά προγράμματα, αλλά και γενικότερα τις παγκόσμιες επιπτώσεις κάποιων από τις τράπεζες αυτές, οι οποίες λειτουργούν κάποιες επαναλαμβάνω από αυτές σε ε, παγκόσμιο επίπεδο. Λοιπόν, αυτή η αξιολόγηση αυτή της ίσης αντιμετώπιση των εμπλεκομένων πώς διασφαλίζεται και διασφαλίστηκε σύμφωνα με τις εμπειρίες τις οποίες έχει συλλέξει μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλώς. Θα ξεκινήσουμε ανάποδα ο κύριος Κάλτον πρώτος. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας σχετικά με την αξιολόγηση των ανταγωνιστικών στρεβλώσεων ή καλύτερα των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού. Ε, είδαμε ότι οι προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπαθούν ε, πράγματι να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις των κρατικών βοηθειών, ενισχύσεων και διαφθρωτικών μέτρων. Όχι μόνο σε σχέση με τις συγκεκριμένες τράπεζες αλλά και με την αγορά συνολικά μέσα στην οποία κινούνται σε κάθε χώρα. Αυτή είναι η υποχρέωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η εμπειρία μου λέγει και γι' αυτή με φωνάξατε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει τη δουλειά της καλά. Δεν υποτιμώ την δυσκολία της συγκεκριμένης αυτής προσπάθειας, ιδιαίτερα όταν σε ένα κράτος μέλος υπάρχουν πολλές τράπεζες που έχουν πάρει κρατικές βοήθειες ενισχύσεις. Συνεπώς είναι δύσκολο να αξιολογήσει κανείς τις συνέπειες αυτής της βοήθειας μεταξύ τους και ανάμεσα σε αυτές και σε τράπεζες που δεν έχουν πάρει βοήθεια σχετικά με την δημιουργία πρωταθλητών της ε, Ευρωομάδας σε σχέση με τις τράπεζες που δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά ίσως θα πρέπει να τα δει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει αν αυτό είναι που τους ενδιαφέρει. Η βασική τους στόχος είναι η σωστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και σωστός ανταγωνισμός ανάμεσα στους κοινοτικούς εταίρους. κύριος Βίνκ. Είπα ότι αυτή η ισότιμη αντιμετώπιση των εμπλεκομένων στην αγορά είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και αναφέρθηκα ήδη σε αυτό. Ακούσα και τον κύριο Αλμούνια να λέει ότι θέλουμε να καταργήσουμε το κατώτερο αυτό πλαίσιο και να καταστήσουμε πιο αυστηρό το πλαίσιο, εν πάση περιπτώσει, μέσα στο οποίο θα κινηθούν τα πιστοτικά ιδρύματα. Πράγματι αυτό το όριο που έχει καθοριστεί μέχρι τώρα είναι σχετικά αφαίρετο, αλλά παρόλα αυτά έχει σημασία να διασφαλιστεί η ισότιμη αντιμετώπιση των ε, ιδρυμάτων και εφόσον καταργηθεί, δεν θα πρέπει να καταργηθεί μόνο για νέες αιτήσει κρατικής βοήθειας ενίσχυσης, αλλά και για αυτές οι οποίες έχουν τύχει βοήθεια στο 2008 και 2009. Υπάρχουν πάρα πολλές τράπεζες που ήταν λίγο κάτω από το όριο αυτό, το 1,9 ας πούμε, και αν αλλάξει το πλαίσιο η αλλαγή αυτή θα πρέπει να ισχύσει για όλες τις τράπεζες χωρίς διακρίσεις. Υπήρξαν ορισμένε συζητήσει σε σχέση με την βοήθεια ρευστότητα από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είπα ότι το ισότιμο αυτό πεδίο αντιμετώπισης δεν λαμβάνει μόνο την ανακεφαλαι... τις προσπάθειες ενίσχυσης σε νέα κεφάλαια, αλλά γενικότερα τις παρεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όταν μια τράπεζα δεν πάει καλά, είτε πηγαίνει άσχημα και ε, προχωράει σε πτώχευση λόγω ρευστότητας, είτε λόγω έλλειψης κεφαλαίων. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί να μην λαμβάνεται υπόψη η ρευστότητα στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, και να μην λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα παρέμβαση τη Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Α πούμε ότι τώρα μπορεί να δανειστεί κανεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με 1% και να τα διαθέσει στην αγορά δανείων με 4%. Υπάρχει δηλαδή ένα περιθώριο εδώ 3% χωρί καμία προφανή προσπάθεια για να πετύχει κανεί. Αυτή η διαφορά δεν είναι κρατική ενίσχυση. Από πλευρά Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα κατανοώ ότι έχουν αναλάβει τις δικές τους ευθύνε και βλέπουν τα πράγματα με τον δικό τους τρόπο, αλλά ενιολογικά αυτό είναι κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνω πώς δεν λαμβάνεται υπόψη σοβαρά. Τέλος είναι πάρα πολύ δύσκολο να φέρει κανείς σε σύγκληση τα ευρωπαϊκά και τα αμερικανικά πρότυπα. Αυτό βλέπει όμως τα τελευταία χρόνια ότι μια επιχείρηση σαν την ING η οποία λειτουργούσε και στις Ηνωμένε Πολιτείες, δεν μπόρεσε να ωφεληθεί από το αμερικανικό προγράμματα. Ενώ οι αμερικανικές τράπεζες που ωφελήθηκαν από το πρόγραμμα αυτό μπορεί να λειτουργούν στην Ευρώπη χωρίς κανένα πρόβλημα και να ανταγωνίζονται τις ευρωπαϊκές ε, τράπεζες οι οποίες και αυτές πήραν ή δεν πήραν κρατική βοήθεια. Υπάρχει μια αναντιστοιχία δηλαδή εδώ στο τι συμβαίνει στο στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με την ερώτηση ότι η ισότιμη μεταχείριση είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Όσον αφορά τις εγγυήσει, όπως είπα και προηγουμένως, ένα σημαντικό βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση ελήφθη με τις αποφάσεις που άρχισαν να ισχύουν από τον Ιούλιο ότι οι τιμές των εγγύσεων αυξήθηκαν και συνδέθηκαν με την αξιοπιστία των τραπεζών. Επίσης, θα υπάρχει αναθεώρηση βιωσιμότητας, το οποίο αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό και θα μειώσει, νομίζω, σε σημαντικό βαθμό τις τρευλώσεις στον τομέα των εγγύσεων. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, κύριος Πέρες Ρενοβάλες. Ευχαριστώ. Εφόσον μιλούμε για ισότιμη μεταχείριση, θα ήθελα να πω ότι είναι σημαντικό δεν μιλάμε μόνο για τις ε, κρατικές εγγύησεις. Όταν, για παράδειγμα, ένα μέρισμα δεν εξυπηρετείται για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της μη εξυπηρέτησης των δανείων, και αν δεν υπάρχουν περιορισμοί καθόλου μετά την ε, λήψη κρατικής ενίσχυσης, αυτό δημιουργεί προβλήματα μεταξύ των μετόχων ε, και δεν δημιουργεί καθόλου θεμητό ανταγωνισμό και ούτε ισότιμη μεταχείριση. Όσον αφορά την ε, στρατηγική εξόδου, δεν πρέπει να μας διαφεύγει ότι όταν μιλάμε για ένα ίδρυμα που δεν είναι βιώσιμο και λαμβάνει κρατική ενίσχυση, αυτό επηρεάζει την εμπιστοσύνη σε ολόκληρο το σύστημα, γιατί δεν υπάρχει εμπιστοσύνη και συνεπώς τα μετά υπάρχουν προβλήματα ρευστότητας, γιατί υπάρχει έλλειψη εμπιστοσύνης ε, στις ε, τράπεζες. Ευχαριστώ. Ε, thank you. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Συνεχίζουμε με τις ερωτήσεις των συναδέλφων και αν έχουμε λίγο χρόνο στο τέλος ε, θα δώσω το λόγο και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί μπορεί να θέλει και εκείνη να απαντήσει σε κάποιες ε, ερωτήσεις αλλά δεν μπορώ να σας δώσω το λόγο πάνω από μία φορά. Ο Χωσέ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι το δεύτερο αυτό τμήμα της ακρόασης μας είναι πολύ πιο χρήσιμο, διαπιστώνω. Ειδικότερα στην άσκηση του λειτουργήματός μας ως ε, νομοθετών. Αναφέρεται το γεγονός ε, ότι δεν ήταν καλή ανάλυση. Θα είναι καλή ανάλυση όταν θα μπορούμε να αξιολογήσουμε ολόκληρο το σύστημα των μέτρων τη Ευρωπαϊκή ε, Κεντρική Τράπεζα αλλά και των κρατικών ενισχύσεων. Και διαπιστώνω επίση ότι οι εκπρόσωποι του τομέα διαπιστώνουν σοβαρέ στρεβλώσει ανταγωνισμού. Για παράδειγμα, μιλήσαμε για την ε, εξόφληση των ενισχύσεων αυτών και μας ε, είπατε ότι εξαρτάται από τις διαστάσεις, ε, από το μέγεθος των, τραπεζών, όπως επίσης και από το εθνικό σύστημα, κάτι το οποίο βέβαια αντίκειται στην ουδετερότητα της οποίας υποτίθεται ότι είναι εγγυητής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μα είπατε επίσης ότι δεν υπήρξε ισότητα, ότι υπήρχαν ενισχύσεις ε, για ιδρύματα που δεν έλαβαν ε, ενισχύσεις ε, γιατί αντιμετώπιζαν προβλήματα ρευστότητας και θα έπρεπε να διαλυθούν ουσιαστικά για να μην δημιουργηθούν προβλήματα σε ολόκληρο το σύστημα. Υπάρχει το θέμα της ασφάλειας δικαίου από τη μία, αλλά από την άλλη υπάρχει και το εξής ζήτημα τι μπορούμε να κάνουμε ώστε από εδώ και στο εξή να μην υπάρχουν στρεβλώσεις ε, ανταγωνισμού, ώστε οι τράπεζε που δεν σεβάστηκαν την αρχή αυτή να μην ευνοηθούν στο μέλλον. Πώς θα κάνουμε λοιπόν, πώς θα γίνει ώστε να, να, να, να διορθωθεί αυτό, αυτή η κατάσταση. Είπατε ότι είστε υπέρ της αναδιάρθρωσης του στήματος, το είπε και ο Επίτροπος Βαρνιέ, για να βοηθηθεί πραγματική οικονομία. Και γιατί αυτές οι ενισχύσεις Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και οι κρατικές ενισχύσεις δεν κατάφεραν να βελτιώσουν ε, την κατάσταση των πιστώσεων και τι θα γίνει προκειμένου να υπάρξει ε, αύξηση των πιστώσεων. Ευχαριστώ. Από την άλλη μεριά αυτή τη φορά θα αρχίσουμε. Αντίστροφα, ο κύριος Ρενοβάλες. Θα απαντήσω ισπανικά. Ε, στον κύριο Μαργκάγια. Λοιπόν, για τα μέτρα για την αποφυγή των στρεβλώσεων. Νομίζω ότι απλώς θα πρέπει να εφαρμόσουμε σωστά αυτά τα οποία είχαμε στην ανακοίνωση της Επιτροπής, ε, διότι εδώ έχουμε μία περίπτωση ε, όπου όπου υπάρχουν πολλές τράπεζες στην αγορά και ε, χρειάστηκε να ε, πουληθούν ορισμένα περιουσιακά στοιχεία. Το θέμα είναι όμως η εφαρμογή και πώς αυτή θα εφαρμοστεί. Το δεύτερο δηλαδή όσον αφορά ε, τη, τη δυνατότητα των πιστώσεων, εάν ε, κοιτάξετε ακριβώς το τι γίνεται, θα δείτε ότι κατά τα τελευταία χρόνια ε, εκτός από ορισμένε εξαιρέσεις οι τράπεζες που δεν βοηθήθηκαν ήταν αυτές οι οποίες μπόρεσαν περισσότερο να καλύψουν τα έξοδα των επιχειρήσεων και να δώσουν δάνεια προς τους πολίτες. Ο κύριος Λεβί. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Καταρχήν κύριος Βίνκ μάλλον, με συγχωρείτε, ε, ήδη αναφέρθηκε επανειλημμένος ε, από τους προηγούμενους ομιλητές ότι πρέπει να έχουμε μία προσεκτική προσέγγιση, διότι πρέπει να τελειώσουν οι κρατικές ενισχύσεις, αλλά προσεκτικά, χωρίς να γίνουν ε, πωλήσει της πυρκαγιάς, διότι αυτό δεν θα βοηθήσει κανέναν. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει υπάρχει κίνητρο για ε, να τελειώσει αυτό το σύστημα και αυτό αναφέρθηκε και από προηγούμενους ομιλητές. Δηλαδή όχι ε, ε, μία ποινή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν προσπαθείς να ξεπληρώσεις την κρατική βοήθεια αλλά ένα σύστημα αποπληρωμής των κρατικών ενισχύσεων. Αυτό ήταν το μόνο το οποίο ήθελα να προσθέσω. Ωραία. Λοιπόν, τώρα ερχόμαστε στην, στον Άντωνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τέσσερις ερωτήσεις. Μία για κάθε ομιλητή. Ε, ο κύριος Μπέσσερντερ Δενό Βάλες αναφερθήκατε σε πέντε θέματα όσο αναφορά την αναθέτηση ε, ε, θεώρηση, τη μεταρρύθμιση. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε πώς ε, σκοπεύετε να ε, διεκπαιρεώσετε και να διαχειριστείτε την κρίση. Κύριε Βίνκ, ε, αναφερθήκατε στις διεθνείς κρατικές ενισχύσεις. Μιλάτε για τις δυνατότητες δυνατότητες ε, βοηθείας ε, για την έξοδο από την κρίση. Αναλόγως των περιοχών στην Ιαπωνία, στην Ευρώπη, στην Ασία υπάρχουν ε, διαφορετικές αποδόσεις. Επίσης κύριε Λεβί είπατε ότι καλό θα ήταν να παρατείνουμε αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή εσείς πώς αντιλαμβάνεστε την ε, βαθμία διέξοδο από αυτό το σύστημα βοηθειών και ενισχύσεων. Ο κύριος κάρτον αναφέρθηκε ε, εις την ε, ανάγκη μέτρων και ε, κάποιος άλλος αναφέρθηκε στην προβλεψιμότητα. Πώς θα υπάρχει διακριτικότης και προβλεψιμότητα. Οπότε, οι ίδιες ερωτήσεις με τη, στην αντίστοιχη σειρά απαντήσεως. Όσον αφορά τα διάφορα θέματα, θα ήθελα να σας πω ότι οι μηχανισμοί εποπτείας και η διακυβέρνηση των επιχειρήσεων είναι το θέμα που μας απασχολεί, διότι τα προβλήματα πάντοτε είναι συνδεδεμένα με κίνδυνους, διότι προασπίζουμε ένα πρότυπο όπου η διαχείριση των κινδύνων είναι στο προσκήνιο. Δηλαδή ε, γι' αυτό και το πρόγραμμα της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι ένα σωστό πρότυπο το οποίο θα έπρεπε να ακολουθήσουμε. Όσον αφορά το μηχανισμό εποπτείας, πολλές φορές είπαμε ότι αυτό το οποίο απέτυχε δεν ήταν τόσο ε, το σύστημα το ρυθμιστικό όσο ή το εποπτικό. Το, μιλήσαμε για το ισπανικό σύστημα το οποίο είναι πολύ πολύ κοντά στις ε, επιχειρήσεις και όπου υπάρχει ένας ε, μηχανισμός ε, επεμβάσεως που επιτρέπει να επεμβαίνουμε πριν εκδηλωθεί η κρίση τουλάχιστον πριν υπάρξουν επιπτώσεις στην εθνική οικονομία και κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προλάβουμε άλλες κρίσεις. Επανερχόμενος ε, στην ερώτησή σας για τις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών. Πιστεύω ότι οι μεγάλες διεθνείς τράπεζες συμβάλλουν στην διεθνή οικονομία και αυτό επιβεβαιώθηκε στην, σε μια πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου διότι μπορούν να αναπτύξουν νέες ε, υπηρεσίες, μπορούν να διαφοροποιήσουν τη δυνατότητά τους να ε, εξυπηρετήσουν και τις πολυεθνικές εταιρείε σε πολυεθνικό επίπεδο και έχουν μία ε, πρόσθετη, ε, προστιθέμενη αξία από πλευράς ανταγωνισμού επίσης. Οπότε πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στον κατακαιρματισμό τέτοιων τραπεζών. Χρειαζόμαστε και στο μέλλον ε, ε, στην διεθνή αγορά να υπάρχουν ε, μεγάλοι παίκτες και εάν να μειώσει η Ευρώπη αυτούς τους παίκτες της θα αποδυναμώσει και την οικονομία της. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αναθεωρήσουμε τις κρατικές ενισχύσεις που παρέχονται στις τράπεζες αλλά η μακροοικονομική επίπτωση θα πρέπει επίσης να αξιολογηθεί κατά περίπτωση δηλαδή δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο την επίσημη νομική σκοπιά αλλά και τις επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Ένα από τα σημαντικά θέματα το οποίο έγινε αντικείμενο ε, θα έλεγα λήψης μέτρων ήταν η αξιολόγηση των εγγύσεων. Αυτό το οποίο είδαμε εμείς στην έρευνά μας είναι ότι οι τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Ένωση πλήρωσαν τα ίδια τέλη θα έλεγα για τις εγγυήσεις αυτές ανεξαρτήτως χώρας και ανεξαρτήτως αξιολόγησης πιστοτικού ιδρύματος. Κανονικά ο μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας θα έπρεπε να λάβει υπόψη την αξιολόγηση και τη βαθμολόγηση του πιστοτικού ιδρύματος, αλλά για διάφορους λόγους οι τράπεζες, οι περισσότερες από αυτές, πλήρωσαν από 80 με 120%, ε, ε, με 120%, με 120 μάλλον. Αυτό ήταν το κόστος των εγγυήσεων. Χώρες όπως τώρα η Ιταλία, η Πορτογαλία και η Ισπανία είχαν φυσικά το ίδιο κόστος ασφάλισης αλλά ταυτόχρονα πλήρωσαν υψηλότερα ποσά από ότι οι γερμανικές τράπεζες. Αλλά το κόστος έκδοσης των ομολόγων ήταν πολύ χαμηλότερο γιατί στην ουσία έγιναν αυτόματα συγκρίσεις με το γερμανικό χρέος. Λοιπόν, αυτό δημιουργεί μερικές μορφές τρέβλωσης και έχει νομίζω διορθωθεί εν πολλής από τα μέτρα τα οποία υιοθετήθηκαν τον μήνα Ιούλιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια άλλη στρέβλωση η οποία και αυτή έχει μειωθεί πολύ αφορά την ποιότητα αυτών ε, οι οποίοι θα έλεγα τη ζήτηση για δάνεια. Τους τελευταίους 12 μήνες είδαμε ότι η αξιολόγηση πιστοληπτική των τραπεζών που ζήτησαν τέτοιες εγγυήσεις από τα μέσα του 2009 μειώθηκε κατά πολύ. Στην ουσία λοιπόν είχαν υψηλότερο πιστοληπτικό κίνδυνο. Αυτό σημαίνει ότι οι αδύναμες τράπεζες παραμένουν εξαρτημένες από τις εγγυήσεις αυτές και στη δεύτερη περίοδο της κρίσης και γι' αυτό οι αποφάσεις οι οποίες λήφθηκαν τον Μάιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν σωστές. Γιατί θα πρέπει να υπάρξουν ε, εκθέσεις βιωσιμότητας πριν ζητήσουν περαιτέρω εγγυήσεις και πριν ανοίξουν το ρομπινέ για να πάρουν τη βρύση, για να πάρουν τα χρήματα που περιμένουν πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν να τα επιστρέψουν. Τώρα σχετικά το πώς μπορώ να συνδυάσω την ευελιξία και τη διακριτικότητα από τη μία με τον έλεγχο των λογιστικών στοιχείων και, την, και τον, γενικά και τον έλεγχο της ποιότητας των πιστοτικών ιδρυμάτων από την άλλη. Κοιτάξτε, εμείς αντιμετωπίζουμε κάθε παρέμβαση κατά περίπτωση. Από την άλλη οι συζητήσει στις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Μπαρνιέ σε σχέση με τον έλεγχο των λογιστικών των πιστοτικών ιδρυμάτων έχουν σαν στόχο την δημιουργία ενός νέου πλαισίου που θα αφορά το σύνολο των ιδρυμάτων που συμμετέχουν στην αγορά. Υπάρχει λοιπόν μια διαφορετική θα έλεγα συζήτηση εδώ. Θα ήθελε κάποιο μέλος να επανέλθει λοιπόν σε ερωτήσεις. Όχι, σε αυτή την περίπτωση θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν ξέρω ποιος θα πάρει το λόγο της Ευρωπαϊκής, από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σχρήμαν από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα ήθελα να σχολιάσω τις παρατηρήσεις του κυρίου Πέρες για την άνηση μεταχείριση την οποία πιθανώς αντιμετωπίσαμε τις διαφορετικές παρεμβάσεις στο τομέα των κρατικών ενισχύσεων. Εμείς δεν εξετάσαμε μόνο τη μεμονωμένη κατάσταση σε κάθε χώρα αλλά και κάθε περίπτωση σε κάθε χώρα αλλά και γενικότερα τις ανάγκες για ε, σταθερότητα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ανάλυση βέβαια της αντίδρασης δείχνει ότι θα πρέπει ε, να ε, είναι ανάλογη με την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά μέσα στην οποία λειτουργεί η τράπεζα η οποία παίρνει τα χρήματα. Προσπαθούμε εμείς να διασφαλίσουμε ισότιμες συνθήκες έτσι ώστε να οφήσουμε προς την απαραίτητη μεταρρύθμιση και τελικά μόνο βιώσιμες επιχειρήσεις θα παραμείνουν όρθιες στο τέλος. Αυτό σημαίνει σωστή κατανομή των πιστώσεων, αυτό σημαίνει ότι οι ίδιες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμμετέχουν επαρκώς και γαλύπτοντας το κόστος της μεταρρύθμισης και θα ήθελα να μάθω ποιες ήταν οι επιχειρήσεις οι πιστοτικές οι οποίες πήραν βοήθεια από πλευράς μας και οι οποίες ταυτόχρονα έδωσαν και υψηλό μέρισμα στους μετόχους τους. Αυτό θα ήθελα να μας ενημερώσετε. Εν πάση περιπτώσει ε, η προσπάθεια της μεταρρύθμισης εσωτερική έγινε και από την προσπάθεια εκποίησης κάποιων περιουσιακών στοιχείων ή ε, τμήματων, εκχώρησης τμήματων του ενεργητικού συγκεκριμένων πιστοτικών ιδρυμάτων και ταυτόχρονα υπάρχουν και κάποια επιμέρους ε, μέτρα. Uh, υπάρχουν επίσης και οι περιορισμοί με το λεγόμενο price leadership ban, δηλαδή ε, να μην ωφελούνται ε, και να μην μπορούν να προτείνουν προϊόντα οι τράπεζες που παίρνουν τις βοήθειες αυτές ε, τα οποία δεν μπορούν να προσφέρουν στην αγορά οι τράπεζες που δεν έχουν τύχει τις ίδιες βοήθειες. Νομίζω ότι υπήρξαν περιπτώσεις αρνητικές σε επίπεδο εθνικής αντιμετώπισης και στις Ηνωμένε Πολιτείες. Ξέρετε τι έγινε με την Lehman Brothers ήταν ε, πολύ σοβαρή η περίπτωση αυτού, η πολιτική ήταν ε, ότι θα μπορούσε να υπάρξει μια μετα, περίοδος μεταρρύθμισης, αναδιάρθρωσης που θα μπορούσε όμως να οδηγήσει και στην πτώχευση και τη ρευστοποίηση του ενεργητικού της συγκεκριμένης τράπεζας. Υπήρξαν ορισμένες περιπτώσεις και μπορεί να υπάρξουν και άλλες όπου η τελική απόφαση ε, θα είναι να κλείσει το πιστοτικό ίδρυμα αλλά όχι στα πλαίσια μιας άγριας πτώχευσης η οποία θα δημιουργούσε πολλές δυνατότητες κατάχρησης. Το χρηματοπιστωτικό σύστημα στην Ευρώπη δεν κατέρευσε όπως έγινε στις Ηνωμένε Πολιτείες. Πράγματι ε, είναι φυσικό να αντιμετωπίζει κανείς τις τράπεζες οι οποίες βοηθήθηκαν πιο αυστηρά από τις υπόλοιπες. Η ING έχει ξεπεράσει το 2%, έχει τύχει υψηλών ποσοτήτων βοήθειας και ενίσχυσης. Τα μέτρα αυτά βοήθησαν την ING να παραμείνει στην αγορά να συνεχίσει να είναι κυρίαρχη η θέση της και υπήρξαν ε, επίσημα παράπονα από πλευράς των ανταγωνισμών σας λόγω της επιθετικής σας πολιτικής σε ορισμένες ε, εθνικές αγορές. Χωρίς την κρατική βοήθεια η οποία δόθηκε όχι από μια θα έλεγα αμερικανική εταιρεία αλλά από τον Ολλανδό φορολογούμενο συγκεκριμένη περίπτωση συνεχίσατε ε, να λειτουργείτε. Συμφωνώ επίσης μαζί σας με το Price Leadership Ban Πράγματι αυτή ε, είναι μία αρχή η οποία ε, δημιουργεί προβλήματα στις βασικές αρχές λειτουργίας του ανταγωνισμού. Πρέπει να είναι κανείς ικανός να ανταγωνίζεται ακόμα και με τη βοήθεια την οποία έχει πάρει από την κυβέρνηση. Η Ολλανδική αγορά είναι μια πολύ συγκεντρωτική αγορά θέλω να πω ότι ε, ζητήσαμε, αν, ζη, ζητήσαμε την δυνατότητα αυτή να την αλλάξει η ING σημαίνει ότι δεν θα υπάρχει ε, ε, κανένα πρόβλημα στην Ολλανδική αγορά. Και αν η ING δεν ήταν διατεθειμένη να αλλάξει τις υποχρεώσεις που είχε αναλάβει, τότε δεν θα μπορούσαμε και εμείς να αλλάξουμε την ε, δυνατότητα επιβολής του Price Leadership Ban. Εμείς κάνουμε αναλύσεις επί τη βάση του προγράμματος αναδιάρθρωσης, το οποίο υποβάλλεται από το κράτος μέλος και από την επιχείρηση, την πιστοτική, την εταιρεία την πιστοτική και με την συγκεκριμένη έκθεση βιωσιμότητας ε, να μπορεί να ζήσει δηλαδή στην αγορά η πιστοτική αυτή εταιρεία χωρίς ε, να την χάνει κρατικής εγγύησης και βοήθειας να συμμετέχει η ίδια η επιχείρηση στο κόστος της αναδιάρθρωσης της εσωτερικής και να μην υπάρχουν στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό. Αν το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης το οποίο μας υποβάλλεται από τα κράτη-μέλη και το οποίο γίνεται αντικείμενο επεξεργασίας με βοήθεια από την ίδια την εταιρεία και αν καταλήξουμε σε μια κάποια συμφωνία λοιπόν τότε θα υπάρξει μια τελική απόφαση. Εμείς δεν αποφασίζουμε για τα προγράμματα αναδιάφρασης μόνοι μας σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι λίγο περίεργο να ισχυρίζεται κανείς ότι μπορεί να υποβληθεί ένα πρόγραμμα, να μας υποβάλλεται ένα πρόγραμμα, να εγκρίνουμε το πρόγραμμα και μετά να μας πηγαίνετε στα δικαστήρια. Εν δεν θέλω να μιλήσω περισσότερο γι' αυτό γιατί η διαδικασία είναι δικαστικά ανοιχτή ακόμα. Uh, Υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία συνδέονται με την δικαστική αυτή διαδικασία στα οποία δεν μπορώ να αναφερθώ. Παρ' όλα αυτά διευκρινίσαμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι υπέρ της πρόορης αποπληρωμής αυτό ε, θα μπορούσα, θα θέλαμε να ισχύσει και στην περίπτωση του ING, αλλά θέλουμε η όροι αυτή της αποπληρωμής ε, να είναι οι σωστοί. Αν εγώ χρωστώ ε, κάτι σε κάποιον και πρέπει να πληρώσω κάτι επιπλέον για τη δανείστηκα, αν τα δώσω τα χρήματα νωρίτερα και θεωρηθεί ότι επειδή τα δίνω νωρίτερα δεν θα πληρώσω το επιπλέον ποσό, αυτό είναι ένα πρόβλημα. Είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί. Τώρα για την απαλλαγή από συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία, από ενεργητικά τμήματα του ενεργητικού κτλ. Νομίζω ότι η περίοδος αυτή για το λεγόμενο divesting μπορεί να είναι μεγαλύτερη χρονικά από αυτή η οποία έχει συζητηθεί μέχρι τώρα οι αποεπενδύσεις αυτές μερικές φορές ε, δημιουργούν πρόβλημα γιατί οι επιχειρήσεις οι οποίες προβαίνουν σε τέτοιου είδους ενέργειες τις κοστολογούν σε ένα επίπεδο το οποίο εμείς δεν βρίσκουμε ότι είναι πράγματι τόσο υψηλό. Θα πρέπει να υπάρξει συν σαν παράδειγμα ένα τμήμα ε, της επιχείρησης το οποίο θα πρέπει να φύγει, πρέπει να απολυθεί διότι ε, δεν βοηθάει την επιβίωση της επιχείρησης ή πρέπει να απολυθεί για να μπορέσει να αποπληρωθεί το χρέος προς το δημόσιο ενωρίτερα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους μπορεί να υπάρξει μια τέτοια διάθεση στην αγορά τμήματων των επιχειρήσεων και τέτοιου είδους ενέργειες βοήθησαν και ανταγωνιστές να μπουν σε μια αγορά στην οποία όμως παραμένει η επιχείρηση συγκεκριμένη λόγω ακριβώς της κρατικής βοήθειας για τα θέματα της διαφάνειας, τα οποία αναφέρθηκε και ο κ. Σκάλτον. Εμείς δημοσιεύουμε όλες τις αποφάσεις μας και το κάνουμε το ταχύτερο δυνατόν και εξαρτώμεθα και από την ιδιωτική πλευρά να μας πει τι μπορούμε να δημοσιεύσουμε ακριβώς και θα πρέπει να συμφωνήσουμε με την εταιρεία ε, ε, για το τι μπορούμε να δημοσιεύσουμε και τι δεν μπορούμε να δημοσιεύσουμε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λειτουργεί με διαφάνεια στον συγκεκριμένο τομέα της δημοσίευσης των στοιχείων και όλα αυτά θα τα βρείτε σε επίπεδο λεπτομεριακό στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Για το 2% τώρα. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε γιατί βάλαμε το όριο αυτό του 2%. Το 2% που ήταν κατά κάποιο τρόπο το καταφύγιο στο οποίο μπορεί να προσφύγει κανείς για να προχωρήσει στα προγράμματα αναδιάρθρωσης, είχε τεθεί στο τέλος του 2008 την εποχή που υπήρχε πρόβλημα με τη δανειοδότηση των αναγκών της οικονομίας. Και κάποιες κυβερνήσεις εκείνη την εποχή δεν ήθελαν να δώσουν χρήματα γιατί δεν ήξεραν ακριβώς ποια θα ήταν η κατάληξή τους. Αν θέλουμε τώρα οι επιχειρήσεις να δανείζουν στην πραγματική οικονομία και από την άλλη να απειλούνται γι' αυτό παρότι κάνουν κάτι το οποίο είναι κατεξοχήν υγιές και χρήσιμο τότε είναι ένα πρόβλημα και γι' αυτό είχαμε ορίσει το 2% αλλά δεν είναι πρόβλημα πλέον, υπάρχει δυνατότητα δανεισμού της πραγματικής οικονομίας και μπορούμε να αλλάξουμε τις προϋποθέσεις και τις συνθήκες και δεν έχει καμία σχέση με άνηση μεταχείριση των πιστοτικών ιδρυμάτων μεταξύ τους. Έχει αλλάξει η κατάσταση και μπορούμε να αλλάξουμε πλέον τους κανόνες. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ζητήσω από καθέναν από τους ομιλητές μας, ε, μήπως θέλουν να συνοψίσουν για μερικά λεπτά για οποιοδήποτε θέμα. Δεν θέλουμε να υπησέλθουμε σε πολύ συγκεκριμένες περιπτώσεις για τις δικαστικές υποθέσεις, την αναδιάρθρωση. Είναι γεγονός. Υπάρχει μια δυνατότητα δικαστικής προσφυγής αν κάποια εταιρεία θεωρείται θεωρεί ότι έχει τύχει, ότι έχει τύχει άνησης μεταχείρισης. και υποθέτω ότι πάνω από μία τράπεζες βρίσκονται σε αυτή τη θέση. Περιμένουμε να δούμε ποιο έχει δίκιο και ποιο έχει άδικο. Δεν ε, σημαίνει, δεν, δεν ε, μπορεί κανείς ε, να απαγορεύσει στις τράπεζες ή στις εταιρείες να ακολουθήσουν αυτήν την οδό απλώς και μόνο επειδή υπήρχαν αυτά τα προγράμματα αναδιάρθρωσης. Δεν ξέρω, δεν λέω ότι πρέπει υποχρεωτικά να πάρετε το λόγο, αλλά αν θέλετε να συνοψίσετε, ευχαρίστε. Ναι, ένα σημείο μόνο θα ήθελα να θέσω, λέει ο κύριος Κάλτον. Αυτά που άκουσα και από τα μέλη του πάνελ αλλά και από τους ευρωβουλευτές, πραγματικά Βλέπω όρεξη για καλύτερο απολογισμό ή καλύτερη διαφάνεια από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όχι μόνο για συγκεκριμένες αποφάσεις, όχι τόσο για τα στοιχεία της κάθε απόφασης, αλλά πώς γίνεται να συγκεράσουμε τις διάφορες ε, περιπτώσεις, να υπάρχει μια ακαιρεότητα του συστήματος και επίσης πώς προσπάθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη διάρκεια της ε, ε, κρίσης αυτής να αναλύσει τις συνθήκες στις διάφορες τράπεζες των διαφόρων κρατών μελών ε, και πώς ελήφθησαν μεμονωμένες αποφάσεις σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Ε, είναι πάρα πολύ δύσκολο το εγχείρημα αυτό και νομίζω ότι η διαφάνεια είναι πολύ σημαντική. Θέλω να κάνω μια πιο, ένα πιο γενικό σχόλιο και συμφωνώ ότι δεν πρέπει να ε, υπησερχόμαστε σε λεπτομέρειες. Δεν είμαστε στις Βρυξέλλες, όχι στο Λουξεμβούργο και πιστεύω ότι κάθε Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να εφεσιβάλει. Εν πάση περιπτώσει οι τράπεζες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη πολλών πολιτών και ουσιαστικά η τραπεζική λειτουργία βασίζεται στην εμπιστοσύνη. Εάν δεν έχετε την εμπιστοσύνη των πελατών σας, των καταθέτων και των υπαλλήλων, υπάρχει πρόβλημα. Οπότε το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι να επανακτήσουν την εμπιστοσύνη των ε, καταναλωτών, ε, της κοινωνίας, των ε, υπαλλήλων τους και νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει επίσης να αναφέρουμε. Άλλωστε συμφωνώ με την άποψη του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι η οι τράπεζες δεν πρέπει να αναλαμβάνουν υπερβολικούς κινδύνους οπότε ε, έχουμε ε, συμφωνήσει ε, σε ένα ποσοστό κερδών και ήδη τον πρώτο χρόνο αποπληρώσαμε το ίμιση της βοηθείας στο Ολλανδικό κράτος αυτό είναι το μόνο που θα είχα να σας πω όσον αφορά την συγκεκριμένη τράπεζα. Εγώ θα ήθελα να σας πω ότι, όπως είπαμε και προηγουμένως, τα περισσότερα μέτρα για να αποκαταστήσουν τον ανταγωνισμό πρέπει να συμμορφώνονται στις αποφάσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρέπει λοιπόν να εφαρμόζονται σωστά και για μένα είναι πολύ δύσκολο να βρω μία πραγματική ισορροπία ανάμεσα στις διάφορες πτυχές αυτού του θέματος για να δω πώς μπορούμε να διατηρήσουμε τον ανταγωνισμό αφενός και να έχουμε ε, βιώσει μεσοντότητες που να επιβιώσουν ε, και αυτό το αντιμετωπίζει και η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η οποία λέγει ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να αξιολογηθεί η βιωσιμότητα για να δούμε εάν ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε. Και το θέμα αυτό έχει πολλές ε, επιπτώσεις. Αυτό που θα ήθελα λοιπόν να προσπαθήσω να πω είναι ότι σαν ε, εταιρεία θα πρέπει εφόσον ε, συμμετέχουμε σε διαδικασίες και αγοράζουμε ε, χρεόγραφα από διάφορες ε, ε, εταιρείες που αντιμετωπίζουν πρόβλημα να ε, έχουμε ένα επίπεδο ισότητος μεταξύ μας. Ευχαριστώ. Θα ήθελα εδώ να ολοκληρώσουμε αυτή την ακρόαση, να πω ότι ευχαριστώ τους πάντες. Θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ορισμένα από τα κείμενα των παρουσιάσεων διατίθενται και θα υπάρχουν στην ισοσελίδα και άλλα θα συμπληρωθούν με ε, σκέψεις που βασίζονται σε όσα ελέγχθησαν και ε, όποιος θέλει να κάνει κάτι τέτοιο ή αν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να μας στείλει άλλα στοιχεία για τους ευρωβουλευτές θα είμαστε ευγνώμονες. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Έχουμε άλλο ένα θέμα στην ημερήσια διάταξή μας αλλά πρώτα πρέπει να επιτρέψουμε στους ομιλητές να αποχωρήσουν. Okay, now the final item on the agenda. Λοιπόν, το τελευταίο θέμα της ημερησίας διατάξεώς μας είναι το θέμα 12 σχετικά με τις, ε, ε, τον κανονισμό του Συμβουλίου σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις που διευκολύνουν την ε, πάυση λειτουργίας μη ανταγωνιστικών αθαγορυχίων. Δυστυχώς δεν θα μπορέσει να παρίσταται ο κύριος Ραπκάη αλλά το ενημερωθήκαμε μόνο αφού είχε τοποθετηθεί το θέμα αυτό στην ημερησία διάταξη. Άρα δεν θα υπάρξει εισαγωγή από τον κύριο Κάι. δεν έχει αναθέσει και σε κάποιον άλλο να κάνει την εισαγωγή ανταυτού. Οπότε Φίλιπ, όποιος άλλος θέλει να αναφερθεί σε αυτό είναι στη διάθεσή του. Απλούστατα ε, θέλει κάποιος να σχολιάσει αυτό το θέμα. Όλοι φεύγουν, οπότε... Ε, άνοιξα και έκλεισα τη συζήτηση. Εδώ έχουμε ε, ένα, ε, μία προθεσμία για τις τροπολογίες ε, και θα συζητηθεί εννέα... Νοεμβρίου στην Επιτροπή ε, για να μπορέσει στην Ολομέλη να συζητηθεί ή στην δεύτερη Ολομέλεια του Νοεμβρίου. Ε, ο ένας από τους λόγους ήταν ότι δεν είχαμε τις μεταφράσεις. Όταν θα υπάρξουν οι μεταφράσεις θα υπάρξει και η επαναφορά στην ημερήσια διάταξη και έτσι ο καθένας θα μπορέσει να ενημερωθεί για την τύχη των τροπολογιών του. Η επόμενη συνεδρίασή είναι Δευτέρα 18 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο και λύεται η συνεδρίαση.